Dear uh, welcome to you all uh, uh, this evening um, to this. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην κοινή συνάντηση των, της συνεδρίας αυτής. Ο κύριος Γκουαλτιέρη θα προεδρεύσει σε αυτή τη συνεδρίαση. Καλώς ορίζουμε τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης και τους Επιτρόπους Τάισεν και Μοσκοβισή για αυτόν τον οικονομικό διάλογο, για την οικονομική επισκόπηση για την ανάπτυξη, για το μηχανισμό προειδοποίησης. Συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η συνάντηση εντάσσεται στο πακέτο διαλόγου είναι το πρώτο βήμα αυτού του ετήσιου κύκλου. Πρώτα ξεκινάει ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν οι καθήλυνα αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και το Κοινοβούλιο περάσει στον οικονομικό διάλογο και δώσει δυνατότητα στους εισηγητές και σε όλους σας την ε, ευκαιρία να συζητήσετε την ε, ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη την ετήσια έκθεση για την απασχόληση, να συζητήσετε με την Κομισιόν, να λογοδοτήσει σε εσά η Κομισιόν, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Θα δώσουμε καταρχάς το λόγο στους επιτρόπους μας που θα μιλήσουν ο ένας μετά τον άλλον για 20 λεπτά. Και εν συνεχεία θα έχουμε δύο γύρους ομιλητών, στο πρώτο τμήμα και στο δεύτερο τμήμα που θα αναλάβει να προεδρεύσει η Αντιπρόεδρος Βουλσκό, θα έχουμε τρεις γύρους ομιλητών Καταρχάς, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης για την εισαγωγή του. Mr. Chair, ε, Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, με τα χαρά σας να σας παρουσιάσω τη δέσμη μέτρων του φθινοπόρου που ξεκίνησε το εξάμεινο, το, θα ξεκινήσει το εξάμεινο το 2017 για την όλη διαδικασία. Θέλουμε μια οικονομική ανάκαμψη. Το ΑΕΠ έχει φτάσει ψηλότερα από ό,τι στα προηγούμενα στις προηγούμενες φάσεις της κρίσης και πρόκειται να αυξηθεί και άλλο του χρόνου. Ιδίω με τι ε, θέσει εργασία που δημιουργούνται, πέφτει η ανεργία τα ποσοστά τη. Οι επενδύσει ε, αυξάνονται ο μέσος όρος του δημοσίου χρέους και η αναλογία ΑΕΠ και δημοσίου χρέους θα συνεχίσει να μειώνεται τα επόμενα δύο χρόνια. Πέραν όμως αυτών που είναι κάπως ενθαρρυντικά, αυτά τα κάπως θετικά σημάδια ε, περιστοιχίζονται και από άλλα αρνητικά. Δηλαδή είναι ευάλωτο το σύστημα ακόμα και οι προοπτικές ε, αύξησης είναι αβέβαιες καθώς υπάρχουν κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις Ιδίω όσο η ανεργία δεν καταπολεμάται πλήρω. Είναι ακόμα σε ψηλά επίπεδα. Η αύξηση και οι ανισότητε του εισοδήματο παραμένουν μεταξύ των περισσότερων χωρών. Το, δημοτικό, το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέο παραμένουν υψηλά και είναι σε πολλές χώρες ε, τα δάνεια που δεν αποδίδουν ε, και πλήττουν τον τραπεζικό τομέα. το συμπέρασμα ότι θα πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπαθίες μας για να στρίξουμε την αύξηση, να προωθήσουμε τις επενδύσεις, να γίνουν απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και να υπάρχουν υπεύθυνε δημοσιονομικές πολιτικές. Για το σκοπό αυτό έχουμε επικεντρωθεί στην κοινωνική δικαιοσύνη και την περισσότερη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Πρώτα απ' όλα για τις ψηλότερες επενδύσεις. Εδώ χρειάζεται η στήριξη της ζήτησης ε, και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να δώσουμε πλήρη εκδίπλωση στο δυναμικό μας. Γι' αυτό που να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και να δούμε τα όρια που υπάρχουν για τις επενδύσεις προς στιγμή, να προωθήσουμε την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση των Κεφαλαιοαγορών, καθώς και ε, τη στήριξη κάποιων εθνικών τραπεζικών τομέων. Επίσης πρέπει να συνεχίσουμε με την ε, υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Στατικικού Επενδυτικού Ταμείου. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας λοιπόν και για, την, ε, για τις επενδύσεις και για τη στήριξη των εισοδημάτων. Στην ε, στρατηγική της νέας αγοράς θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Χρειάζονται φιλόδοξες ε, μεταρρυθμίσεις σε όλα τα κράτη-μέλη. Το ίδιο και υπεύθυνε δημοσιονομικές πολιτικές, που είναι σημαντικέ για τη μακροοικονομική σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μια καινοτομία τη δέσμη μέτρων τη φετινή είναι η δημοσιονομική νέα στάση στην ε, Ευρωζώνη μετά την ομιλία του Πρόεδρου Γιούνκερ. Η ανακοίνωση τη Επιτροπή μιλάει για το δημοσιονομικό προσανατολισμό και για μια σωστή ανάμειξη πολιτικών στην Ευρωζώνη. Πρέπει να υπάρχει σεβασμό των δημοσιονομικών μα κανόνων και να, λάβετε, ε, να λαμβάνετε υπόψη η σταθερότητα του γενικότερου συστήματος. Θα πρέπει προσπάθειες των κρατών μελών να επιδιώξουν τη μακροοικονομική σταθερότητα της Ευρωζώνης με ξυγχρονισμένη ε, ανάπτυξη σε πολλούς τομείς ε, για τη δημοσιονομική πολιτική. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί το ε, υπέρμετρο έλλειμμα καθώς και οι μεσοπρόθεσμοι δημοσιονομικοί στόχοι να επιτυγχάνονται. Θα πρέπει τα επίπεδα που έχουν τεθεί ως στόχοι να ε, επιδειχθούν και να επιτευχθούν. Επίσης, κάποιοι θα πρέπει να στηρίξουν τους δημοσιονομικούς τους προσανατολισμούς μέσω πρόθεσμα, εφόσον μπορεί να χρειαστεί να έχουν περισσότερο εκτατική ε, δημοσιονομική πολιτική, κυρίω στηρίζοντας τι επενδύσει. Θα πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα των ε, κρατικών δημοσιονομικών, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στι δαπάνε, την προτεραιότητα στις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που να στηρίζουν την αηφορία ε, μακροπρόθεσμα. Στι ε, συστάσει μα για την Ευρωζώνη ε, εντοπίζουμε πέντε τομεί δράση. Πρώτα απ' όλα μεταρρυθμίσει που θα τονώσουν την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα, τη στήριξη των δημοσιονομικών προσανατολισμών, την κοινωνική πολιτική και δικαιοσύνη, τη στήριξη του τραπεζικού τομέα και την ολοκλήρωση τη νομισματική και οικονομική ένωση. Όλα αυτά τα πολιτικά εργαλεία δείχνουν την ανάγκη η πολιτική και η διευθυντική ε, συνιστόσα να συνδυαστούν για να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις και να υπάρχει ανάπτυξη. Το 2017 πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις που μπορούν να φέρουν αύξηση με όλες μας τις δυνατές προσπάθειες. Με την κοινή ε, έκθεση για την αύξηση και τη μελέτη των αγορών εργασία των κρατών μελών, βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη διευθυντικές ε, προκλήσει. Υπάρχουν ακόμη ψηλά ε, ποσοστά ανεργία, ιδίω των νέων, με χαμηλά προσόντα ή προβλήματα στην εκπαίδευση και επίση άτυπη εργασία. Υπάρχει επίση το θέμα των των άσυλων και των προσφύγων που εισραίουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζουν με την, στο επίπεδο τη μεταναστευτική πολιτική. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν τις αναχώρασε τάσει να τι ε, ε, εκπληρώσουν με την εκτέλεση των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν όμω πολλέ ευκαιρίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα διευθυντικά ταμεία και τα επενδυτικά ταμεία, την επένδυση για την Ευρώπη και μόλι εγκριθεί από του συνομοθέτε στο πρόγραμμα στήριξη των διευθυντικών μεταρρυθμίσεων. Οι συνέπειε των μεταρρυθμίσεων πολλέ φορέ χρειάζονται χρόνο μέχρι να γίνουν πραγματικότητα. Όμω όσο περισσότερο συνεχιστούν, τόσο περισσότερο οι χώρε θα αυξάνουν το δυναμικό του για ανάπτυξη και θα αντιμετωπίζουν τι μακροοικονομικέ και δημοσιονομικέ ανισορροπίε. Στα επόμενα βήματα θα πρέπει να ε, καλέσουμε όλα τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν τις ε, μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες και να μην ξεχνάμε ότι πέρσι είχαμε 19 χώρες που έπρεπε να λάβουν κατεπηγόντως μέτρα Τώρα θα δούμε τα ευάλωτα σημεία που παραμένουν αρκετά και σημαντικά. Ε, Κυρίε και κύριοι, μετά την επόμενη φάση των αναχώραση τάσεων την επόμενη άνοιξη, η Επιτροπή θα ειδικοποιήσει το διάλογο με τα κράτη-μέλη και του κοινωνικού εταίρου, προκειμένου να πετύχει μια κοινή συνεννόηση για την επιτυχή υλοποίηση των ε, μεταρρυθμίσεων. Για να προετοιμάσει τα εθνικά προγράμματα με την ετήσια ε, μελέτη ανάπτυξης καλούνται και τα εθνικά κοινοβούλια να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή μαζί με του κοινωνικού εταίρου. Και το Ευρωκοινοβούλιο βεβαίω με τι επαφέ που έχει με τα εθνικά κοινοβούλια μπορεί να διδραματίσει εδώ καθοριστικό ρόλο. Και εμεί επαναλαμβάνουμε την αφοσίωσή μα να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάνω, όλα, πάνω απ' όλα χρειαζόμαστε μια ξεκάθαρη αντίληψη του ποιε είναι οι κοινέ μα προτεραιότητε και οι κοινοί μα στόχοι. Αναμένουμε ανυπομονησία το διάλογο μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Dan het eh, woord aan eh, commissaris Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Επίτροπο Τάισεν. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ξεκινώ τονίζοντας ότι βελτιώνοντας αυτά τα οποία αναφέρε ο Αντιπρόεδρος, όλα αυτά που συσχετίζονται με τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιούν τα κράτη-μέλη πρόσφατα για την δυνατότητα ανάκαμψης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Η ανάκαμψη είναι όμως ευάλωτη και δεν ήταν εξίσου αισθητή από όλους τους Ευρωπαίους. Πάνω από 4 εκατομμύρια νέοι βρίσκονται ακόμα χωρίς να έχουν θέση απασχόλησης. 119 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται υπό κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν στη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 25 εκατομμύρια παιδιά μεταξύ αυτών και 23,7% είναι το επίπεδο για ε, εκείνους που ζουν στη φτώχεια υψηλότερο από εκείνο το οποίο ήταν 23,3% του 2009 στην ε, ζώνη ευρώ δεν έχουμε επιστρέψει ακόμα στα επίπεδα 2009 και βρισκόμαστε στα υψηλότερα επίπεδα τα οποία αφορούν την ανάπτυξη και την ανάκαμψη. Παραμένουν αυτά τα προβλήματα λοιπόν κοινωνικά και θέματα φτώχειας. Δεν υπάρχει περιθώριο λοιπόν να είμαστε για αυτοικανοποίηση και η επισκόπηση της ε, τήσιας ανάπτυξης ε, δείχνει πόσο σημαντικές είναι οι τεχνολογικές αλλαγές ε, όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη. Και όπως είπε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας όσον αφορά την κατεύθυνση για την αναπρόθεση της απασχόλησης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με μια υπεύθυνη φορολογική πολιτική ώστε να έχουμε πιο χειροπιαστά αποτελέσματα στην απασχόληση. Θέλουμε επενδύσεις στη γνώση, στην διαβίου εκπαίδευση για να μπορέσει η απασχολησιμότητα να αναπτυχθεί και να μπορέσει η διαφορά μεταξύ υψηλών δεξιοτήτων και μικρότερων δεξιοτήτων να καλυφθεί. Οι δείκτες δείχνουν έλλειψη όσον αφορά τις δεξιότητες ε, του ε, εργατικού πληθυσμού και είναι αναγκαίο λοιπόν να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες οι εργαζόμενοι από βασικές τέτοιες δεξιότητες ε, έως και δεξιότητες και ικανότητες του επιχειρήν Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, αυτά τα μηνύματα στην ετήσια επισκόπηση για την ε, ετήσια ανάπτυξη βρίσκονται και μέσα στο σχέδιο έκθεσης το οποίο δίνει μια επισκόπηση όσον αφορά τις εξελίξεις για τα κοινωνικά θέματα στην Ευρώπη. Το σχέδιο έκθεσης επίσης καταδεικνύει ότι τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη ακολούθησαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην εργασιακή αγορά μεταρρυθμίσεις που συμπεριλαμβάνουν και την δυνατότητα με, για τη δημόσια ε, απασχόληση και δίνοντας ε, και την εγγύηση για τους νέους, για την νεότητα, δίνοντας έτσι ε, μια νέα μορφή στην αγορά εργασίας μειώνοντας όσον αφορά τις ε, μεγάλες διαφορές και αυξάνοντας την αηφορία και την αποτελεσματικότητα των συνταξιδοτικών συστημάτων. Υπάρχει κάποια πρόοδος, αλλά περαιτέρω δράση απαιτείται να αναλυθεί. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να είναι προστατευτικός παράγοντας. Πρέπει να βελτιωθεί το προστατευτικό πλαίσιο από τα κράτη-μέλη μέσα στο πλαίσιο της αγοράς και να αποφευθεί η κοινωνική, ο κοινωνικός αποκλεισμός. Αυτό απαιτεί υποστήριξη στήριξη εισοδημάτων, καθώς επίσης και βοήθεια στην περίθαλψη ηλικιωμένων παιδιών μελών οικογενειών. Περισσότερες προσπάθειες πρέπει να γίνουν για τη συμμετοχή ευρύτερων περισσότερων ανθρώπων στην ε, ε, εργασιακή αγορά. Να υπάρχει ελαστικότητα και επαρκής ασφάλεια. Διάφορα κράτη-μέλη έχουν ήδη αναπτύξει στρατηγικές για την ένταξη μεταναστών με προηγούμενη πείρα και εμπειρία και ένας αριθμός κρατών μελών θα πρέπει να δημιουργήσουν τις επαρκείς δομές ε, για τους μετανάστες ε, και μια στρατηγική πέρα από τις ε, βραχυπρόθεσμες ανάγκες, δίνοντας τη δυνατότητα να διεξαχθεί ένας αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος όσον αφορά τα κοινωνικά θέματα στην αγορά. Πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας κοινωνικές πολιτικές και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον Εν κατακλείδη έχουμε θετικά αποτελέσματα, αλλά περαιτέρω δράση απαιτείται αν θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινωνική αγορά στα εργασιακά. Το ίδιο μήνυμα πρέπει να απευθυνθεί με την ανάγκη υλοποίησης μεταρρυθμίσεων στις αγορές ε, όσον αφορά την Ευρώπη. Περισσότερα πρέπει να γίνουν, αλλά ξεκινάμε ήδη αυτή την ε, δράση υπέρ των πολιτών ε, με την εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων, κυβερνώντων, κυβερνήσεων, ε, πολιτών, κοινωνίας των πολιτών και φυσικά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πράγματι οι δικές σας συνεισφορές και προτάσεις θα έχουν ρόλο κλειδιού. Θα είναι πραγματικά ανεκτήμητες για αυτή την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κ. Μοσκοβισή. Έχετε το λόγο κύριε πίτροπε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές. Με μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάσω μαζί με τους συναδέλφους σήμερα το πακέτο για το φθινόπωρο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ε, βρισκόμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο με πολλέ αβεβαιότητες και όπω ε, εξήγησε και ο Βαλτή, υπάρχει μια οικονομική ανάκαμψη, είναι όμω ευάλωτη, υπάρχει αλλά δεν επιταχύνεται. Ε, αν λάβουμε υπόψη μα τι περιορισμένε προοπτικέ ανάπτυξη στο εξωτερικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν εθαρρύνει τι εξαγωγέ. Ο πληθωρισμό παραμένει ασθενή παρά τις, τα μέτρα οικονομική πολιτική ανεπροηγουμένου. Το ποσοστό ανεργία είναι ψηλό, 10% ε, το είπε και συνάδελφο, ε, και υπάρχει μια μεγάλη υποχρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού στην αγορά εργασία, που φαίνεται κιόλα και με όρου κεφαλαίου. Υπάρχει μια ανάκαμψη των επενδύσεων, αλλά είναι ασθενή, ε, εμποδίζεται από τις ασθενεί οικονομικέ προοπτικές. Υπάρχει ένα πραγματικό κίνδυνο, αυτή η υποχρησιμοποίηση του παραγωγικού δυναμικού ή υποχρησιμοποίηση να γίνει χρόνια και να επηρεάσει την ανάκαμψη. Μέσα από την εξέταση της, της ανάπτυξης του 2017, η Κομισιόν ε, καλεί τα κράτη-μέλη να διπλασιάσουν τις προσπάθειες αυτού που αποκαλεί ε, του τριγώνου της αρετής τη οικονομική πολιτική. Να ξαναρχίσουν οι επενδύσει, να συνεχιστούν διαρθρωτικέ ε, μεταρρυθμίσει και να γίνουν οι απαραίτητε δημοσιονομικέ πολιτικέ. Θα πρέπει τώρα να αναπτυχθούν τα δημοσιονομικά μέτρα, ούτω ώστε να εξισορροπήσουμε τον πόληξη μίξη τη Ευρωζώνη για να υποστηρίξουμε την νομισματική πολιτική τη ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ε, που ήδη κάνει ό,τι μπορεί. Καταρχά, θα πρέπει να υλοποιηθούν 100% οι δημοσιονομικέ απαιτήσει που αφορούν την κάθε χώρα ε, και παρά το γεγονός ε, ότι η οικονομική κατάσταση απαιτεί μια δημοσιονομική πολιτική σχετικά επεκτατική, οι συγκεκριμένες συστάσεις θα οδηγούσαν ε, συνολικά σε μια δημοσιονομική κατάσταση, ένα δημοσιονομικό προσανατολισμό σχετικά περιοριστικό στην Ευρωζώνη, και το 2018. Αυτή η συνολική δημοσιονομική κατάσταση, ο δημοσιονομικό προσανατολισμό, κρύβει μια άνηση κατανομή μεταξύ των κρατών μέλων Αντίθετα από αυτό που θα απαιτούσε ε, μια χρηστή οικονομική διαχείριση για την Ευρωζώνη. Η κατάσταση είναι παράδοξη. Αυτοί που έχουν δημοσιονομικό περιθώριο θέλουν, που δεν έχουν δημοσιονομικό περιθώριο, θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Αυτοί που έχουν δεν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Είναι μια ε, συνολική προσέγγιση που δεν είναι σωστή και απαιτείται μια προσπάθεια για να γίνουν και να βελτιωθούν τα δημόσια οικονομικά και να γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις και οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Η έκθεση για το μηχανισμό επαγρύπνησης εντοπίζει τα κράτη-μέλη για τα οποία θα πρέπει να γίνει η ενδελεχής εξέταση, ε, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο των εκθέσεων αναχώρα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, για να αξιολογήσουμε αν υπάρχουν κάποιες χώρες οι ε, οποίες έχουν μακροοικονομικέ ανισορροπίε που απαιτούν διορθωτικά μέτρα. Η οριζόντια ανάλυση τη έκθεση αυτή για το 2017 δείχνει ότι οι βασικέ πηγέ κινδύνου παραμένουν ουσιαστικά οι ίδιε με αυτέ που εντοπίστηκαν στην έκθεση του 2016. Ό,τι αφορά τι εξωτερικέ ανισορροπίε, ο, ο προσανατολισμό, η προσαρμογή του ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών των χωρών που είναι οφειλέτε ε, μοιάζει να έχει ολοκληρωθεί, αλλά ορισμένε χώρε πιστωτέ εξακολουθούν να έχουν ένα πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών πολύ υψηλό. Αυτή η συμμετρία τη διόρθωση των ανισορροπιών του ισοζυγίου τρεχουσών πληρωμών ε, επιμένει και δημιουργεί προβλήματα οι Τράπεζε έχουν αυξήσει την κεφαλαιοποίησή του και η αντίστασή του στα σοκ γενικά έχει βελτιωθεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διάφορε προκλήσει. Εν κατακλείδη, η έκθεση για τον μηχανισμό επαγρύπνωσης του 2017 δείχνει ότι οι εντελεχείς εξετάσει είναι απαραίτητε για 13 χώρε, 6 λιγότερε από πέρυσι. Αυτέ οι 13 χώρε ήδη είχαν υποβληθεί σε εξέταση στον προηγούμενο κύκλο και είχαν εντοπιστεί διάφορες ανισορροπίες και αυτή, αυτή η νέα εξέταση θα αποτελέσει την αναλυτική βάση για να διατυπωθούν συγκεκριμένες ε, συστάσεις στα πλαίσια της διαδικασίας για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και θα αξιολογηθούν και οι πρόοδο που έχει σημειωθεί από αυτέ τι χώρε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ολοκληρώσω αυτή την παρουσίαση με τι συστάσει για την Ευρωζώνη. Από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο του 2015, οι συστάσεις για την Ευρωζώνη δημοσιεύονται στην αρχή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με την ετήσια εξέταση για την ανάπτυξη. Αυτή η αλλαγή παρακολουθεί τη φιλοσοφία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ούτω ώστε οι κοινέ προκλήσεις να λυθούν υπόψη και αυτό να μεταφραστεί σε ειδικέ συστάσεις αναχώρα το Μάιο. Αυτό έχει δώσει δικαπούς με μια ουσιαστική, ένα ουσιαστικό εμπλουτισμό των συζητήσεων για τι προκλήσει στην Ευρωζώνη. Οι συστάσει, οι ειδικέ συστάσει τη Ευρωζώνη, ε, συγκεντρώνονται στην καλή λειτουργία τη Ευρωζώνη. Η πρώτη σύσταση αφορά τη συνέχιση των πολιτικών που υποστηρίζουν την οικονομική ανάκαμψη και που προωθούν τη σύγκληση, που διευκολύνουν τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και βελτιώνουν τι ε, δυνατότητε προσαρμογή. Η δεύτερη σύσταση αφορά τη δημοσιονομική πολιτική, κυρίω την ανάγκη για την οποία μίλησα, να υιοθετήσουμε έναν προσανατολισμό πολύ πιο θετικό στη δημοσιονομική πολιτική με σεβασμό του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Συνεχεία, η καλή λειτουργία τη αγορά τη εργασία και του, του δημοσιονομικού, του χρηματοοικονομικού συγγνώμη, τομέα ε, είναι η τρίτη και η τέταρτη σύσταση. Η πέμπτη σύσταση αφορά την ανάγκη να επιταχύνουμε τι προσπάθειε για να συμπληρώσουμε την Οικονομική και Δημοσιονομική Ένωση. Συζήτηση με τα κράτη-μέλη για το περιεχόμενο των συστάσεων και για το πακέτο του φθινοπόρου μέχρι στιγμή ήταν έντονε και παραγωγικέ. Το Eurogroup έδειξε ότι προτιμάει ένα προσανατολισμό ουδέτερο αντί για θετικό. Δεν είναι αυτό που ήθελε και που σύστησε η Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά, όμως, ε, δέχεται την ε, αρχή του fiscal stance, του δημοσιονομικού προσανατολισμού. Αυτή η συζήτηση είναι εξελίξη, δεν θα σταματήσει με αυτή την πρώτη συζήτηση, αυτή την πρώτη προσέγγιση. Αυτός ο διάλογος είναι σημαντικός για να αισθανθούμε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι κοινή υπόθεση και να υιοθετηθούν οι δικέ συστάσει ανά χώρα. Χάρη στου στενού δεσμού με τεχνικά κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ε, μείζον εταίρο για να υποστηρίξουμε την εφαρμογή των προτεραιοτήτων και θέλουμε να εμπλέξουμε πολύ στενά αυτά τα εθνικά κοινοβούλια καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους για την εκπόνηση και την εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων προς το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μου δώσατε να κάνουμε εκ νέου αυτή τη συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Αυτό μας φέρνει σε εσά συνάδελφοι. Ξεκινάμε με τον πρώτο γύρο των ομιλητών, με τους ε, συγκητές πρώτα, τον κύριο Χέκμαρ και την κυρία Τούν. Έχετε τρία λεπτά ο καθένας. Κύριε Χέκμαρ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσά Επίτροπε. Νομίζω εδώ υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να τονίσουμε. Πρώτα απ' όλα την ανάγκη να υπάρχει αναβαθμισμένο επίπεδο δημοσίων οικονομικών στις επενδύσεις και στις ε, διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις. Νομίζω αυτό και ε, τελευταία και από εσά εκτός από άλλους αναφέρθηκε. Αλλά σε σχέση με την επισκόπηση για την ανάπτυξη από πλευρά σας, το γεγονός ότι υπάρχει μια ανάπτυξη αλλά χαμηλού επίπεδου πρέπει να μας προβληματίσει και βασίζεται αυτό στην μοναδική μοναδικού χαρακτήρα νομισματική πολιτική. Θα με ενδιαφέρει να ακούσω από σας σε ποιο βαθμό θα λέγατε ότι η χαμηλή ανάπτυξη όπως την βλέπουμε τώρα εξαρτάται από αυτή την μοναδικού χαρακτήρα η νομισματική πολιτική χαμηλών επιτοκίων. Συζητώντας τα χαμηλά επιτόκια όμως αυτό υπογραμμίζει και ένα άλλο πρόβλημα. Και αυτό είναι ακόμα το ότι το επίπεδο επενδύσεων είναι πάρα πολύ χαμηλό ακόμα. Επίσης και όσον αφορά και τα δημόσια οικονομικά σε σχέση με τις επενδύσεις, το βρίσκω πράγματι προβληματικό και ανησυχητικό ότι παρότι έχουμε μοναδικά χαμηλά επιτόκια σε αυτή τη συγκυρία, τα κράτη-μέλη δεν ήταν σε θέση να μειώσουν τα ελλείμματά τους παρά μόνο περιθωριακά. Και όταν βλέπουμε ότι είναι τόσο, σε τόσο χαμηλά επίπεδα τα επιτόκια σε σχέση με την συγκυρία, τι λέει αυτό για το μέλλον διότι η νομισματική αυτή πολιτική μπορεί να μην είναι τόσο αηφόρος ε, μακροπρόθεσμα στο μέλλον. Και νομίζω ότι γίνεται δεκτό αυτό αυτό τι σημαίνει λοιπόν για το μέλλον το να έχουμε μια τέτοια ε, τάση μειώνοντας ε, όσον αφορά τα ελλείμματα. Αν δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη τα πολύ χαμηλά επιτόκια για να δημιουργήσουν μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές ε, συνδυάζοντας τις δράσεις τους για τη μείωση των ελλημάτων, τότε η πρόκληση θα είναι πολύ μεγαλύτερη στο μέλλον όταν αυξηθούν αυτά τα επιτόκια. Και αυτό όχι μόνο επειδή η νομισματική πολιτική είναι εκείνη που είναι υπεύθυνη, αλλά επειδή έχουμε και το σύμφωνο σταθερότητα το οποίο υπονομεύεται και αμφισβητείται. Ε, διότι στη συνέχεια τι θα δούμε αυτά που είδαμε και στο παρελθόν. Δηλαδή θα αυξηθούν τα επιτόκια και αυτό θα έχει άμεσες επιπτώσεις, αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, αλλά και στην χρηματοοικονομική σταθερότητα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι θα σήμαινε αυτό για την απασχόληση, για τις διαρθρωμένες δομημένες μεταρρυθμίσεις και τα ελλείμματα, αν αναμείνουμε και δεν αναλάβουμε δράση αμέσω σήμερα, ελπίζοντας ότι μπορούμε να ε, επεκταθούμε όσον αφορά την, ε, τα ε, ελλείμματα και να μπορέσουμε έτσι να επιβιώσουμε έστω επεκτείνοντας αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι μια μεταφορική αναφορά. Θα ήταν καλό λοιπόν σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις, διαφρομένες μεταρρυθμίσεις, να μπορέσουμε να προβούμε στις μεταρρυθμίσεις αυτές σε μια περίοδο χαμηλών επιτοκίων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροποι, ευχαριστώ για την παρουσίασή σα. Συνάδελφοι, την περασμένη Τρίτη στην Επιτροπή Απασχόληση Κοινωνικών Υποθέσεων είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση που συντάσσουμε. Ε, σε πρώτη φάση, εγώ και οι συνάδελφοί μου με χαρά ακούσαμε ότι φέτο η έμφαση θα δοθεί στην σημασία του να διασφαλίσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη ώστε να τονώσουμε την περισσότερη και συμμετοχικότερη ε, ανάπτυξη. Για την ανάκαμψη όλων των ευρωπαϊκών οικονομιών και για αυτέ που είναι εργασιακά εντατικέ, χρειάζονται διαφορετικέ μεταρρυθμίσει σε πολλά κράτη-μέλη. Έχουμε καλέ ειδήσει. Κάποιε νέε θέσει εργασία από το 2013, 8 ε, εκατομμύρια, 8,5 ε, το ποσοστό ανεργία και σε 71,1% στην ομάδα 18-24. Ε, Προηγουμένω η ανεργία στην Ευρωζώνη ήταν, μάλλον η στην Ευρωζώνη ήταν 10%. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, παρά τις σημαντικές ε, μικρέ βελτιώσει, δεν είναι βέβαιο ότι θα φτάσουμε τον στόχο του 75% απασχόληση για την Ευρώπη του 2020, όπω καθορίζει αυτή η στρατηγική. Ε, εδώ Φαίνεται να είναι ύψιστη προτεραιότητα αυτή για την Επιτροπή. Όμω, αυτή τη στιγμή επενδύσει, οι ψηφιακέ δεξιότητε, η καταπολέμηση τη άτυπη και αδήλωτη εργασία και ούτω καθεξή, φαίνεται να είναι περί τα έργα, αν δεν υπάρξουν θέσει εργασία. Ε, ο αποτελεσματικότερο τρόπο να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια είναι να δώσουμε στου ανθρώπου ευκαιρία να δουλέψουν. Η δεύτερη ερώτησή μου έχει να κάνει με το ρόλο των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων και Προγραμματών στο, στο πλαίσιο τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θα το εκτιμούσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα ενημέρωνε για το τι θεωρεί ότι είναι τα απαραίτητα βήματα για να έχουμε περισσότερο αποτελεσματική χρήση των εργαλείων που προβλέπουν τα ευρωπαϊκά ιδρύματα και προγράμματα για τη δημιουργία δουλειά. Ενώ ποια, ποιες είναι οι πρώτες περιοχέ προτεραιότητα σε σχέση με τη λειτουργία των ιδρυμάτων και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Επίση, είναι σαφέ ότι χρειαζόμαστε βιώσιμα κοινωνικά συστήματα προστασία στην Ευρώπη. Κοινωνική πρόνοια δηλαδή και λογική φορολογία. Είναι λογικό να φανταζόμαστε ότι οι διαδικασίε ε, γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού και ανάγκη κοινωνική πρόνοια ε, σημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρέ μεταρρυθμίσει στα συστήματα των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι όλα τα κρατη πρέπει να θεσπίσουν τουλάχιστον ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα. Δεν είναι αυτό ο μόνο τρόπο να υπάρχει η δίκαιη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασία. Και τέταρτη ερώτηση, τελευταία και λιγότερο σημαντική. Η ανεργία και η φτώχεια είναι επικίνδυνε όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, μπορεί να υπονομεύσουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ω ε, πολιτικό εγχείρημα οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορούν να είναι σε θέση να δουν την ολοκλήρωση να φέρουν κάποιε αλλαγέ και στην καθημερινότητά του. Είναι αναντήρητο γεγονό ότι η φτώχεια παραμένει σε ψηλά επίπεδα, όπω το είπε και η Επίτροπο Τάισεν μόλι. το γεγονό αυτό ε, εντοπίζεται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κίνδυνο φτώχεια και κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 25%. Με άλλα λόγια, περισσότερο από ένα στου πέντε Ευρωπαίου υποφέρει από το φαινόμενο αυτό. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Ποια είναι τα μέτρα που έχει προβλέψει η Επιτροπή και ποιο είναι το μήνυμα που μπορείτε να αποστείλετε για να πείσετε του Ευρωπαίου ότι χρειάζονται περισσότερη Ευρώπη. Ή τέλο πάντων ότι χρειάζονται ευθύ εξ αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βοηθήσουμε του ανθρώπου να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασία. Καταλαβαίνω ότι η ερώτηση είναι πολύ γενική, αλλά νομίζω ότι εφόσον θέλουμε να δούμε και την επικοινωνιακή μα πολιτική και υπάρχει και η άνοδο του ευρωσκεπτικισμού, ε, βλέπουμε κύματα λαϊκισμού να παρασύρουν όλη την Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Ε, θα έλεγα να μα απαντήσουν όλοι οι επίτροποι συνολικά σε 8 λεπτά. Αν γίνεται, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ντομπρόφσκι. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Για την πρώτη ερώτηση. Για το πώς, δηλαδή, το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε με χαμηλά επιτόκια επηρεάζει τις τρέχουσες μακροοικονομικές πολιτικές. Και τι θα συμβεί εάν γίνει αλλαγή στην νομισματική πολιτική. Αυτό τονίζεται και από την ΕΚ την ίδια. Ότι μόνο με εργαλεία νομισματικής πολιτικής δεν μπορεί να λύσει τα διαφορετικά προβλήματα της οικονομίας. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ε, με σύνεση την περίοδο αυτή για να εφαρμόσουν τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συμμερίζεται απόλυτα και το τονίζει πάρα πολύ στις προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής μας. Εν συνεχεία, για την αξιολόγηση του δημοσιονομικού ε, προσανατολισμού. Λέτε λέμε ότι υπάρχει μόνο οριακή βελτίωση στο συνολικό έλλειμμα των οικονομιών. Από το 2% που είχαμε πέρυσι θα πάει στο 1,8% ε, φέτος και 1,5% του χρόνου το συνολικό έλλειμμα της Ευρωζώνης. Υπάρχει μια ε, σταθερή μείωση του έλλειμματος του προϋπολογισμού. Και του χρόνου μάλιστα περιμένουμε μόνο ένα μέρος, μέλος της Ευρωζώνης το οποίο θα έχει έλλειμμα πάνω από το 3% του ΕΠ. Βλέπουμε λοιπόν ότι και τα κράτη-μέλη βαθμιδών βγαίνουν έξω από το, από το πλαίσιο του υπερβολικού ελλείμματος. Υπ' αυτή την έννοια το μήνυμά μας είναι σημαντικό και είναι επαγρύπνηση. Αυτό τονίζουμε και σε αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο τα, κράτη-μέλη τα οποία έχουν υπερβολικό έλλειμμα, που δεν έχουν φτάσει στους ενδιάμεσους ε, δημοσιονομικούς ε, στόχους, θα πρέπει να συνεχίσουν στο μονοπάτι της δημοσιονομικής προσαρμογής. Και τα κράτη τα οποία έχουν περιθώριο στο δημοσιονομικό τους προσανατολισμό πρέπει να κάνουν περισσότερες επενδύσεις και να τονώσουν έτσι την οικονομία. Φυσικά όλα αυτά συνδέονται άμεσα με κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Καταρχάς, πρέπει να υπάρξει ανάκαμψη ε, με πολλές θέσεις απασχόλησης. Η αξιολόγησή μας σήμερα είναι ότι υπάρχει αύξηση στο ποσοστό απασχόλησης. Αυτό το 75% μέχρι το 2020 πλήρης απασχόληση, απασχόληση είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί. Και σε αυτό το ευρωπαϊκό εξάμεινο μιλάμε για ανάπτυξη χωρίς να αποκλεισμού. Και θα υπάρξει αυτό ε, και στις ειδικέ συστάσεις ε, αναχώρα, αλλά η Μαριάν θα μιλήσει περισσότερο για τα κοινωνικά θέματα. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Θα εστιάσω στις ερωτήσεις κυρίας Τούμς. Καταρχάς, για την απασχόληση και τα νούμερα της απασχόλησης. Και το αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε το στόχο του 75% απασχόληση που συμφωνήσαμε υπό την Ευρώπη 2020. Οι προβλέψεις της Κομισιόν δείχνουν ότι με το 71% που έχουμε πάνω κάτω τώρα αν συνεχίσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε και αν εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη διαθωτικές μεταρρυθμίσεις, αν χρησιμοποιήσουν τα ταμεία κτλ., τότε μπορούμε να φτάσουμε στο 75%. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει ως διαμαγείας. Πρέπει να συνεχίσουμε τις ε, σκληρές προσπάθειες μαζί με τα κράτη-μέλη και να εστιάσουμε στις ευκαιρίες απασχόλησης για γυναίκες κυρίως. Να δούμε επίσης τι γίνεται και με του πιο ηλικιωμένου εργαζόμενου, ούτω ώστε και αυτοί να έχουν ευκαιρίε στην αγορά εργασία. Έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε ακόμα για ανθρώπου με χαμηλά προσόντα που δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν τη θέση του στην αγορά εργασία. Επίση, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε μια πολιτική για την αγορά εργασία ενεργή. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνική προστασία και τα επιδόματα θα πρέπει να συνοδευτούν από τι σωστέ υπηρεσίε και τα σωστά μέτρα ενεργοποίηση. Αυτό αναφέρεται σε ειδικέ συστάσεις αναχώρα, στο εξάμεινο και σε όλες τις συστάσεις που απευθύνουμε στα κράτη-μέλη. Τώρα, θα αρκέσει αυτό. Έχετε, πολύ... Έχετε δίκιο, κυρία Τούμ, ότι δεν δημιουργούνται οι θέσει απασχόλησης από μόνε τους. Απαιτούν σωστέ μακροοικονομικές πολιτικές, απαιτούν επενδύσει. Επίση, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι επιχειρήσεις μας δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Διότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης δεν γίνεται από εμά, πρέπει να έρθει από τον ιδιωτικό κυρίω τομέα. Αν δείτε, όλε τι υπόλοιπε κατευθυντήριε γραμμέ για τι πολιτικέ εστιάζουν για την εμβάθυνση τη ενία αγορά και την κεφαλαιακή Ένωση και τη δημιουργία του σωστού κλίματο για τι επιχειρήσει, ούτω ώστε όλα αυτά να συντελέσουν τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ποιε είναι οι βάσει για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, Φαντάζομαι ότι μιλάτε για το Eurofound στο Δουβλίνο και για το ΣΕΝΤΕΦΟΠ, που είναι υπεύθυνα ιδρύματα και οργανισμοί για την ε, επαγγελματική κατάρτιση. Βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το, την υπηρεσία που βρίσκεται στο Τωρίνο. Εμείς μπορούμε να, συστάσουμε, να συστήσουμε πολιτικές, αλλά χρειαζόμαστε δεδομένα για να βασιστούμε. Και χρειαζόμαστε ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, που ξέρουν τα δεδομένα, και που μπορούν να μας εμπνεύσουν και να δώσουν σάρκα και οστά στις πολιτικές μας. Μιλάμε για τριμερείς οργανώσεις, ε, εμπλέκονται και οι κοινωνικοί εταίροι και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, εκεί στο ΣΕΝΤΕΦΟΠ και στο Eurofound και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερες πολιτικές ε, στην Ευρώπη. Οι οργανισμοί αυτοί δεν δημιουργούν από μόνοι του ε, τι θέσει απασχόληση. Το θέμα είναι εμεί ότι πρέπει να έχουμε αρκετέ πληροφορίε για να φτιάξουμε τι σωστέ πολιτικές, τις καλύτερες δυνατές πολιτικές, χάρη στις σωστές πληροφορίες που θα μας δώσουν αυτοί οι οργανισμοί. Ακούστηκε μια άλλη ερώτηση για το αν είμαστε, είμαστε υπέρ των ελάχιστων κοινωνικών προτύπων στην Ευρώπη. Θέλουμε δίκαιη κοινωνία. Και θέλουμε και να υπάρξει σύγκληση μεταξύ των κρατών μελών. Θέλουμε να υπάρξει βέβαια σύγκληση προς τα πάνω, με αναβάθμιση του βιωτικού επίπεδου. Η πρότασή μας για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, για αυτόν ε, γίνεται μια μεγάλη διαβούλευση και συνεισφέρει σε αυτή τη συζήτηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα και θα λάβουμε υπόψη μας σίγουρα τις συνεισφορές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την έκθεση της κυρίας Ροντρίγκε, που νομίζω ότι μόλις υιοθετήθηκε στην Επιτροπή Απασχόλησης. Περιμένουμε επίσης και ψηφο, την ψηφοφορία στην Ολομέλεια και σίγουρα θα εμπνευστούμε από αυτή την έκθεση. Εν συνεχεία, για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει και στο μέλλον. Φυσικά είναι καθήκον των κρατών μελών πρωτίστως, αλλά προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων να ασχοληθούμε με το θέμα. Ξέρετε ότι για αυτό το πολιετέ πρόγραμμα συμφωνήθηκε τουλάχιστον το 20% των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Ταμείων θα χρησιμοποιηθούν για το θέμα της καταπολέμησης του αποκλεισμού, της φτώχειας. Και τα κράτη-μέλη υπέβαλαν προγράμματα τα οποία δείχνουν ότι πάνω από 25% των χρημάτων των διευθυντικών ταμείων και των επενδυτικών ταμείων θα ε, δαπανηθούν ακριβώς για να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για την ένταξη. Επίσης ε, προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη για να πάρουν τα σωστά βήματα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και να αντιμετωπίσουν όσους ε, ζουν σε φτώχεια. Τώρα για αυτού, γιατί χρειαζόμαστε την Ευρώπη. Γίνονται πάρα πολλέ αλλαγέ. Ε, παγκοσμίω αυτή τη στιγμή και στις κοινωνίε μας και στην αγορά εργασία. Υπάρχει παγκοσμιοποίηση, υπάρχει μια τεχνολογική επανάσταση παράλληλα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι στο μέλλον είμαστε αρκετά δυνατοί και ότι οργανώνουμε τις κοινωνίες μας και τις αγορές εργασίας μας με ένα τέτοιο τρόπο, ούτω ώστε θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε τους στόχους με σεβασμό όμως των αξιών μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν την Ευρώπη για να μας υπερασπιστεί στην παγκόσμια σκηνή, για να υπάρξει αλληλεγγύη και βεβαίως είμαστε έτοιμοι για να συζητήσουμε περισσότερο αυτό το θέμα. Ε, τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μοσκοβισή. Θα είμαι πολύ σύντομος, διότι τα περισσότερα απαντήθηκαν. Ο Βάλντις απάντησε στα περισσότερα από αυτά πρώτα ο κ. Χόκμαρκ. Και να πω ότι εξ ορισμού τα επιτόκια θα ανέβουν. Πόσο και πότε ακριβώς δεν ξέρουμε. Αλλά ελπίζουμε να είναι βιώσιμο το περιβάλλον που θα δημιουργηθεί. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας κάνει να χάσουμε χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε καμία περίπτωση δεν θέλει να χαλαρώσουμε ούτε ως προς τις ε, διαδοτικές μεταρρυθμίσεις, ούτε ως προς τις δημοσιονομικές προσπάθειες. Για τους στόχους της ανάπτυξης πρέπει να θυμίσω ότι το ποσοστό των ελλημάτων είναι 6% το 2010 και τώρα είναι 1,5%. Καλό θα να σταθεροποιηθεί το 2017. Όταν λοιπόν ε, θέλουμε μια δημοσιονομική πολιτική η οποία να αντιμετωπίζει τα πράγματα συνολικά, δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά του συμφώνου σταθερότητα. σα ίσα πρέπει να κατανείμουμε σωστά τι προσπάθειέ μα σε διαφορετικά πεδία μάχη, ιδίω για χώρε που δεν έχουν κάνει προσπάθειε συγγύανση ε, και για όσου ιδίω έχουν και κάποιο περιθώριο ελιγμού. Το πρόβλημα είναι να μην οδηγηθούμε σε αυτό το αντίστροφο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αυτοί που έχουν κάποιο περιθώριο ε, να μην κάνουν αυτά που ζητάμε και να χαλαρώσουν και άλλοι να κάνουν τα αντίθετα. Ευχαριστούμε. Οπότε τώρα περνάμε στο δεύτερο γύρο μιλητών, με 1,5 λεπτό ο καθένα. Ξεκινάμε με την Επιτροπή ΕΜΠΛ, η κυρία Ριμπέιρου, για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπη, καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσω χαιρετώντα την Επιτροπή, διότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στην ανάλυση των προπολογισμών για το 2017 και για το κοινωνικό βάρος ε, του ευρωπαϊκού συστήματος. Όπω ξέρετε, με απασχολεί όλη αυτή η διαδικασία από την αρχή τη θητεία μα το 2014 και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη στην ισορροπία που αναζητούμε μεταξύ τη κοινωνική διάσταση και του σκέλου του οικονομικού. Πρέπει να εξακολουθήσουμε με πολιτικέ όπου οι Ευρωπαίοι πολίτε να κατανοούν, να βλέπουν ότι πραγματικά εργαζόμαστε για, ε, για του ίδιου. Να αισθανθούν ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εργάζονται προ το δικό του συμφέρον. Και υπ' αυτήν την έννοια πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, διότι πρέπει να βρεθεί μια πραγματική ισορροπία μεταξύ των θέσεων των ε, Επιτροπών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Αυτό το σημείο ισορροπίας θα πρέπει να ε, ενέχεται σε κάθε φάση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το ίδιο και για το Συμβούλιο. Πρέπει να ενισχύσουμε και να πείσουμε το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να ενισχύσει το Συμβούλιο των Κοινωνικών Υποθέσεων, το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Επίση, να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να κάνει κάθε δυνατή και ε, ε, βέλτιστη προσπάθεια για να έχουμε πραγματικό διάλογο με του κοινωνικού εταίρου είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο, διότι αυτή είναι μια ε, αναγκαία προπόθεση για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε νέε πολιτικέ. Και είναι και μια ερώτηση που ήθελα να τη θέσω προ του εκπροσώπου τη Επιτροπή. Φέτο αναφέρεται επανειλημμένο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάγκη να επενδύσουμε περισσότερο, διότι μέσω των επενδύσεων θα καταφέρουμε να έχουμε ανάπτυξη. Ήθελα να καταλάβω ποιο είναι το όριο, αυτό είναι το πιο σημαντικό και θα κλείσω, Πρόεδρε. Ε, γιατί υπάρχει το θέμα των προπολογισμών της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Ποια είναι το όριο που χωρίζει τις επενδύσεις που μπορεί να είναι υπερβολικές και το χρέος που μπορεί να είναι υπερβολικό. Διότι οι επενδύσεις είναι καθοριστικές για να υπάρξει ανάπτυξη. Όμως αυτό θα δημιουργήσει χρέος και θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμφώνου. Ευχαριστώ. Αν μπορείτε όλοι να σέβεστε τα χρονικά όρια, ιδάλλως δεν θα μπορέσουν να πάρουν όλοι το λόγο. Τώρα για του σοσιαλιστέ και δημοκρατέ, ο κύριο Περέιρα από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαιρετίζω και εγώ του κύριου επιτρόπου. Η πιο σημαντική καινοτομία των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2017 είναι χωρί αμφιβολία η σύσταση μια πολιτική δημοσιονομική που θα είναι μέτρια επεκτατική Θέλω να καταστήσω σαφές ότι η σοσιαλιστική ομάδα υποστηρίζει στεναρά με κάθε τρόπο αυτόν τον νέο προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως πρέπει να, κατα... να σημειώσουμε κάτι εκφράζοντας τη θλίψη μας για την αντίσταση που αυτός ο προσανατολισμός ε, δημιουργεί από πλευρά κρατών που έχουν μεγαλύτερο περιθώριο δημοσιονομικό και τη ίδιας της Ευρωομάδας. Η συνέπεια αυτού είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι η συνέπεια ότι η ζώνη ευρώ το 2017 υπό την έννοια της ίδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνεχίσει μια λανθασμένη δημοσιονομική πολιτική. Μπορεί να είναι μετριοπαθώς επεκτατική και μπορεί να είναι μετριοπαθώς περιοριστική όμως θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δύο εξή πράγματα. Πρώτον, τι πρωτοβουλίες πολιτικές θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να δημιουργήσει μια πολιτική συνένεση πιο διευρυμένη γύρω από αυτή την δημοσιονομική πολιτική που θα είναι μετριοπαθώς επεκτατική. Δεύτερη ερώτηση που αφορά τους κανόνες και κανονισμούς διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει ένα παράδοξο στους κανόνες και κανονισμούς που ουσιαστικά παρακολύουν να, να ακολουθεί μια ορθή πολιτική δημοσιονομική. Θέλω να ρωτήσω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για να τροποποιηθούν οι κανόνες της δημοσιονομικής πολιτικής ώστε να μπορέσει η πολιτική δημοσιονομική να είναι η ορθότερη και η πιο επιτυχημένη. Ευχαριστώ. Euh, σας είχα ακούσει, συγγνώμη. Πολύ γρήγορα. Για την απασχόληση κυρίως διορτώ για κάποιε μεταρρυθμίσεις. μεταρρυθμίσει. Παραδείγματα θα σα δώσω. Με τα μεταρρυθμίσει στον τομέα τη εργασία. Βλέπουμε ότι αυξάνεται η ευελιξία, αυξάνεται η μη ασφαλή εργασία, δηλαδή η επισφαλής εργασία, οι, μειώνεται ο κοινωνικό διάλογο που καθορίζει και του μισθού. Φτωχαίνουν οι πολίτε. Τι σκέφτεστε γι' αυτό κανονικά όταν αυξάνεται η ευημερία ε, αυξάνεται και η ανάπτυξη. Εδώ πέρα έχουμε το αντίθετο. Είμαστε σε μια αρνητική συγκυρία. Δεύτερο, μας μιλήσατε και τις συντάξεις. Είπατε ότι θα πρέπει να συνδέσουμε τις συντάξεις με το προσδόκιμο ζωής. Και όμως βλέπουμε ότι η απασχολησιμότητα των ε, εργαζομένων άνω των 50 ε, είναι πάρα πολύ χαμηλή, πιο χαμηλή. Επίσης μιλήσατε για το ιδιωτικό πυλώνα της, ε, της σύνταξης, που είναι ο πλέον άνισος σήμερα και ειδικά για τις γυναίκες. Η πρόσβαση στην εργασία. Δεν βλέπω τίποτα για το work-life work balance, δηλαδή για την ισορροπία ζωή, επαγγελματική ζωή και ιδιωτική ζωή. Αν θέλετε να αυξήσετε την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία, θα πρέπει να μιλήσετε γι' αυτό. Κυρία Τάισεν, μιλήσατε για την παγκοσμιοποίηση. Στην έκθεση ή στην ανακοίνωση που δημοσιεύσατε λέτε ότι υπάρχουν 30 ε, εκατομμύρια θέσει απασχόληση που δημιούργησε το διεθνέ εμπόριο, οι εξαγωγέ δηλαδή. Αναφερόμαστε σε απασχ... θέσει απασχόληση που χάθηκαν επίση στο τομεί όπω τα στη σιδηρουργία, ε, που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση. Νομίζω ότι σήμερα στην Ευρώπη ε, πάμε με το κεφάλι κάτω, μουλαρίσια, προς την παγκοσμιοποίηση που δημιουργεί χαμένους, οι οποίοι, για τους οποίους δεν φροντίζει κανένας. Από το ECR. Ο κύριος Μπέντλουκ, ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Η ερώτησή μου απευθύνεται προς την κυρία Τάισεν. Κυρία Τάισεν, σας ευχαριστούμε που αναφερθήκατε στο πρόβλημα της ένταξης ε, των προσφύγων και μεταναστών στα όσα αναφέρατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής αν γίνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντωμεταξύ εδώ και περίπου ένα χρόνο ξέρουμε περίπου πόσοι άνθρωποι με ποιες δεξιότητες έρχονται και ήρθαν σε εμά. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε καν πώς ε, η δυνατότητα ολοκλήρωσης και ε, αφομοίωσης των αγορών, εργασιακών αγορών για τέτοιους ανθρώπους που έρχονται σε εμά με πολύ λίγες και χαμηλές δεξιότητες. Δηλαδή ποιες ε, εργασιακές αγορές βλέπετε να έχουν το μεγαλύτερο δυναμικό για ανθρώπους που βοηθητικά θα μπορούσαν να δράσουν στις οικοδομές, στη γεωργία ή θα μπορούσαν να προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες και μπορούν να προσφέρουν ε, μη εκπαιδευμένες ε, δεξιότητες, μη ε, ασκημένες δεξιότητες. Θα ήθελα να γνωρίζω ποιο είναι το αποτέλεσμα αν τα εξετάσατε αυτά. Αν δεν τα εξετάσατε να μάθω γιατί δεν εξετάσατε αυτή την προοπτική. Διότι η κατανομή προσφύγων και μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως δημιουργήθηκε πρόσφατα δεν διευκολύνει σίγουρα την δυνατότητα ένταξης αυτών στις αγορές εργασία και μάλιστα υπό άλλε προϋποθέσεις. Αν συμβαίνει λοιπόν έτσι το ότι η κατανομή αυτών των προσφύγων και μεταναστών δεν ανταποκρίνεται στι δυνατότητε ε, απορρόφησής του από τι αγορέ, θα ήθελα να γνωρίζω τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την ελευθερία κυκλοφορία αυτών των ανθρώπων, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν εκεί που θα έχουν τη δυνατότητα ή την απλούστερη δυνατότητα που θα του διανοίγεται να βρουν απασχόληση. Και τέλο θα ήθελα μου πείτε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετείται στον ελάχιστο μισθό. Αν τον ελάχιστο μισθό τον θεωρεί πρόσκομα στην ολοκλήρωση και ένταξη αυτών των εργαζομένων ή αν το θεωρεί ως προστασία αυτών των εργαζομένων. Ευχαριστώ. Και τώρα, η Επίτροπη για δύο με τρία λεφτά ο καθένας, σας παρακαλώ, όχι παραπάνω, γιατί υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, που να μιλήσουν όλοι. Ε, θα επικεντρωθώ στις ερωτήσεις που αφορούν το δημοσιονομικό προσανατολισμό και τους δημοσιονομικούς κανόνες και στα θέματα που συνδέονται με τις επενδύσεις. Καταρχάς, για το ερώτημα που ακούστηκε για το δημοσιονομικό προσανατολισμό, το συμπέρασμα του Eurogroup του Ιουλίου Μίλησε για ένα συνολικό ε, ουδέτερο ε, δημοσιονομικό προσανατολισμό. Και το ΕΚΟΦΗΝ θα επανέλθει στο θέμα αυτό τον Ιανουάριο. Η Κομισιόν συνεργάζεται με το Συμβούλιο για την πρότασή μας που κάναμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το Δημοσιονομικό Προσανατολισμό. Για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στις αρχές του τη περσινή χρονιάς εμείς εκδώσαμε μία ανακοίνωση για την καλύτερη χρήση της ευελιξίας με σεβασμό των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και ανάπτυξη. Υπάρχει ε, επαρκή ευελιξία ε, που εμπεριέχεται στου ε, ισχύοντες κανόνε και θα πρέπει να σεβαστούμε αυτούς τους κανόνες, να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία, αλλά δεν σκοπεύουμε να, και επομένως δεν σκοπεύουμε να προτείνουμε αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη, αλλά θέλουμε να απλουστευτούν οι κανόνε. Πρόσφατα υπάρχει μια, φτάσαμε σε μια συμφωνία για μεγαλύτερη ε, χρήση των όρων αναφορά για τι δαπάνε, ούτω ώστε να βλέπουμε τι δημοσιονομικέ επιδόσει των κρατών μελών. Για το θέμα των επενδύσεων. Οι επενδύσει είναι μία από τι προτεραιότητε τη Κομισιόν. Αυτό το τονίζει το επενδυτικό σχέδιο και για την Ευρώπη και η αποτελεσματική χρήση του, ε, ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και των επενδυτικών ταμείων που είναι στα κράτη-μέλη προτεραιότητα για μας. Υπάρχει όμως και το θέμα της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ειδικά αν υπάρχει υπερβολικό έλλειμμα στα κράτη-μέλη ή υπάρχει υπερβολικό δημόσιο Δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς βιώσιμα και διατηρήσιμα δημόσια οικονομικά. Θα πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία λοιπόν ανάμεσα στις, στη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη και σε μία μακρόπνοη ε, δημοσιονομική βιωσιμότητα. Από την αρχή της θητείας μας εμείς θέσαμε μεγάλη έμφαση στην μεγαλύτερη εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σε διάφορες φάσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου και θα συνεχίσουμε να τους εμπλέκουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τάισον. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να, είμαι, να, να, να συντομεύσω αυτή τη φορά. Θέλω να ευχαριστήσω Ριμπέρο για το γεγονός της παρέμβασης αυτής και το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο ικανοποιείται για τη διαδικασία αυτή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που έχει πιο κοινωνικό χαρακτήρα. Το κάναμε αυτό και εμένα και συνεργαζόμαστε φυσικά με τους υπουργούς στο υπουργικό επίπεδο. Για το ρόλο ΕΣΚΟ πρέπει να αποφασιστεί αυτό φυσικά από τους υπουργούς ε, σε σχέση με τα θέματα ΕΣΚΟ και τα άλλα οικονομικά θέματα όσον αφορά τις ε, ε, δικαιοδοσίες τους. Γιατί την κυρία Ρένα για το θέμα των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων και το τι πρέπει, ποια θα είναι η έκβαση όλων αυτών σε σχέση με τους όρους ε, απασχόλησης και εργασίας ε, ή τη φτώχεια των εργαζόμενων λόγω των προτύπων στην αγορά εργασίας και υπάρχει η ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη αποδεκτικότητα, αποδοχή. Από τη μία πλευρά πρέπει να γίνει αυτό, από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη ασφάλεια όμως ως αντιστάθμισμα. Και σίγουρα όσο περισσ, όσες περισσότερες αλλαγές θα γίνονται κατά τη διάρκεια του βίου των ανθρώπων θα πρέπει στη μεταβατική περίοδο να υπάρχει μια προσφορά υπηρεσιών ώστε οι πολίτες να μπορούν τις ανάγκες τους να τις καλύπτουν όσον αφορά την ποιότητα ζωής τους. Έγινε και το ερώτημα για την ποιότητα ζωής και την ισορροπία των συντελεστών αυτής της ζωής. Καθώς γνωρίζετε όλες αυτές οι συνοδευτικές προτάσεις που αποσύρθηκαν. Υπάρχει όμως μια νέα πρόταση που βρίσκεται υπό εκπόνηση αυτή τη στιγμή και βρίσκεται στο πρόγραμμα εργασίας μας για το 2017. Χωρίς αμφιβολία θα έχουμε ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά του χρόνου, το 2017, για τις συντάξεις και ε, ε, την προσαρμογή στο προσδόκιμο ζωής ε, είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε να το εξετάζουμε. Πρέπει οι σύνταξεις να είναι αηφόρες και πρέπει να εργάζονται επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι για να μπορέσουν να καταστούν αηφόρες οι συντάξεις. Πρέπει να υπάρχει επάρκεια κάλυψης και να δούμε αν θα είναι δυνατόν να διασφαλιστεί ένα επίπεδο ζωής, ένα επίπεδο ευημερίας για τους συνταξιοδοτούμενους Πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι εργαζόμενοι όμως που θα συνεισφέρουν με τις εισφορές τους για να διασφαλιστεί αυτό το επίπεδο ευημερίας των συνταξιούχων. Και μετά για την ερώτηση του κυρίου Λούκε όσον αφορά τους πρόσφυγες και μετανάστες εγώ έκανα λόγο για πρόσφυγες κυρίως. Ε, τα δύο τελευταία χρόνια πολλούς ε, ε, μετανάστες έχουμε δεχτεί στις χώρες μας και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ενταχθούν στις οικονομίες και στις χώρες μας. Θέλουμε να βελτιωθεί η κατάστασή τους, να δοθούν ευκαιρίες σε αυτούς τους ανθρώπους, να προσφερθούν ευκαιρίες να βρουν θέση απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Είναι ο καλύτερος τρόπος να ενταχθούν στην κοινωνική και οικονομική ζωή των χωρών μας. Να δούμε τι θα γίνει όμως στις αγορές εργασίες, Δεν το, δεν το, δεν το γνωρίζουμε επακριβώ. Παρακολουθούμε όμως εκ του σύνεγγυ τα πράγματα να δούμε πώς εξελίσσονται και ποιες τάσεις ακολουθούνται. Καθώς επίσης ε, και τη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου διότι ένα ποσοστό αυτών των κονδυλίων αφορά ακριβώς την καταπολέμηση του αποκλεισμού και την ένταξη στην κοινωνία και στην οικονομία των πολιτών. Τώρα, τι πρέπει να γίνει σε σχέση με την αγορά εργασίας. Πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση των ανθρώπων που προσέρχονται σε εμά, να ταυτοποιηθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητές τους και το δυνατόν γοργότερα να μπορέσουν οι κυβερνητικές υπηρεσίες να τους ε, ε, συνδράμουν για την εξέβρεση θέσης, ε, θέσεως απασχόλησης. Να βοηθηθούν επίσης όσον αφορά τις γλωσσικές γνώσεις τους, την εκμάθηση μιας γλώσσας. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν σε ένα αηφόρο επίπεδο και όλα αυτά να συσχετίζονται και με το επίπεδο παραγωγικότητας και δημιουργικότητας. Όπως γνωρίζετε τα θέματα του ελάχιστου μισθού ή όχι και για το πώς αυτά όλα συνδιαμορφώνουν ε, το πλαίσιο ε, το οικονομικό. Αυτά δεν είναι όμως αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι αρμοδιότητες των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν ε, αυτό πρέπει να δούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα πιο αποτελεσματικά. Και πάλι πολύ σύντομα γιατί οι απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί. Η Επιτροπή θα εμείνει θα μείνει στον αγώνα της για να καταστήσει κατανοητή το πόσο η συναθρισμένη δημοσιονομική συμβολή είναι μία σκέψη εύστοχη. Έχουμε παραμείνει στο Eurogroup στα συμπεράσματα του περασμένου Ιουλίου. Όμως η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι αυτή η εξέταση θα πρέπει να γίνεται συστηματικά. Γιατί οι περισσότεροι είναι πεπισμένοι για το πόσο είναι σκόπιμα αυτά τα μέτρα. Εγώ, όπω και ο Κερούν Ντάισεμπλουμ, έχω την αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεταβατική. Θα υπάρχουν όλο και περισσότερα, χάρη στην επιτυχία του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη, χώρε που θα έχουν περισσότερο περιθώριο λιγμών και θα μπορούν να το αξιοποιήσουν με τρόπο θετικό. Αυτό θα μα επιτρέψει να αποφύγουμε να επικεντρωνόμαστε σε μια ή δύο χώρες κάθε φορά, απλώς γιατί το απαιτεί περίσταση. Ευχαριστούμε, Επίτροπη, για το δεύτερο μέρος αυτής της συζήτησης. Και τώρα ο λόγος στην συνάδελφο. Κυρία Ούλσκοφ, ευχαριστώ για το δεύτερο μέρος λοιπόν αυτής της συζήτησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τις αναχώρασεις τάσεις. Εάν δούμε την υλοποίηση των αναχώρασης τάσεων, το 2012 ήταν μόνο 11%. Βεβαίως, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό ήδη, αλλά χειροτερεύουν τα πράγματα. Το 2015 είναι μόλις 4% πλήρως ε, εκτελεσμένων και υλοποιημένων συστάσεων. 52% καθόλου υλοποίηση και 44% λιγάκι περίπου. Είναι πολλά αυτά που μπορεί να σημαίνει αυτό το εν μέρη, καθόλου και λίγο. Φαντάζομαι ότι θα αισθάνεστε όλοι μεγάλη απογοήτευση γι' αυτό και σα δημιουργεί ματέωση. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν για να αντιμετωπίσετε αυτή την τάση, την ε, φθήνουσα και να αυξηθούν αυτά τα ποσοστά, διότι ιδάλω κανεί δεν φαίνεται να τα παίρνει σοβαρά τι αναχώρε τάσει και δεν δείχνει να υπάρχει πρόθεση να τι πάρει. Ευχαριστούμε κύριο Γκέργε από του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Έχετε το λόγο αξιότιμη επίτροπη, κυρία Τάισαν, για την δική μου ομάδα μπορούμε να σας πούμε σε σχέση με την υποστήριξη από το Ευρωκοινοβούλιο της ε, προσέγγισης ε, του τριγώνου επενδύσεων υπεύθυνη ε, δράσης και σωστής, σωστών δαπανών. Έχουμε ήδη παρκώς παρουσιάσει όλα αυτά. Δύο ερωτήσεις παρακαλώ. Αν δει κανείς στην Ευρώπη τι γίνεται, θα δει ότι Πολλές φορές οι σημαντικές ε, διαθροτικές μεταρρυθμίσεις δεν προχωρούν. Ούτε καν ξεκινούν πολλές φορές. Είναι καλή η βάση αυτή, ώστε ήδη τώρα να μιλάμε για μια διεύρυνση του ΕΦΣΥ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, νέου. Ή μήπω υπάρχουν ε, κυβερνήσεις ε, που θέλουν ε, να αποσυμφορηθούν απλώς μέσω αυτών των δράσεων. Δεν είναι αυτό αντιπαραγωγικό. Η, δική, η η εννοια την οποία έχετε εκπονήσει είναι ρεαλιστική. Για παράδειγμα, μια χώρα όταν χρειάζεται χρειάζεται χρήματα. Όταν όμως πολλές μεταρρυθμίσεις, σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε ένα δημοψήφισμα έχουν απορριφθεί και στη Γαλλία φαίνεται ότι επίκαιρα ε, ε, σε αυτή τη συγκυρία δεν εγκρίνονται όλα αυτά. Έχει ένα ε, πρόγραμμα αναδίπλωσης Plan B η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ιδέες για να αντιμετωπιστεί η αποτυχία τέτοιων κυβερνήσεων και για τα χρήματα σε σχέση με τα οποία, τα οποία θα πετηθούν ε, για την ε, σύγκληση όσον αφορά αυτά τα κράτη. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιέγκας από την ΚΟΕ. Τρία λεπτά, γιατί μιλάτε εκ μέρους και των δύο επιτροπών. Ευχαριστώ πολύ. Μία πρώτη παρατήρηση, διότι είμαι σε απορία. Αφού στην Πορτογαλία, ως γνωστόν, μετά από την αλλαγή συσκεπισμού δυνάμεων στην πολιτική, στο πολιτικό προσκήνιο, η κυβέρνησή μας φέτος έκανε τα πάντα ανάποδα από ό,τι ζητούσαν οι συστάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών. Άφηξε τον ελάχιστο μισθό, ε, μείωσε τις αμοιβές, ε, ανέστηλε τις ιδιωτικοποίησεις, ε, θανάσιμο μάρτυμα και περιέργως το έλλειμμα βελτιώθηκε. Η οικονομία αυξήθηκε. Ξεπέρασε τις ε, προβλέψεις του, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κυρίως τις προβλέψεις της ίδιας της κυβέρνησης. Ω προ την ε, ανάπτυξη λοιπόν και την κατάσταση τη πορτογαλική οικονομία, να ε, σημειώσουμε ότι παρόλο που η ανάπτυξη αυτή παραμένει αδύναμη και έφταστη, ωστόσο μια ερμηνεία πιο σφαιρική υποδεικνύει ότι η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στη συνεισφορά των εξογωγών σε ρευστό, περίπου 60 δις ευρώ, της εσωτερικής κατανάλωσης περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, αλλά κυρίως στην ε, στα 150 εκατομμύρια επενδύσεων που είχαν αρνητικέ, αρνητικό αντίβαρο. Δηλαδή πέφτουν οι επενδύσεις. Αυτό ήταν ε, κυρίως κάτι που παρατηρήσαμε στο τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς. Γι' αυτό λοιπόν ήθελα να με εξηγήσετε εσείς τι απάντηση δίνετε σε αυτή την κατάσταση. Τι απόκριση μπορείτε να, δώσετε ώστε η Ένωση των Κεφαλαγορών, το πρόγραμμα Juncker, η Τραπεζική Ένωση είναι οι κλασικέ συνταγέ, αυτέ που επιβάλλονται εδώ και 10 χρόνια και που δεν έφεραν καμία λύση. Καμία λύση για την πορτογαλική οικονομία. Καμία σωτηρία. Και μια άλλη πτυχή που έχει να κάνει με την ενεργεία και έχει περισσότερο με την απασχόληση να κάνουν όλα αυτά. 30% ενεργεία των νέων. Τι απάντηση έχουμε μετά από το σύνολο των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ε, υλοποιηθεί ανά την Ευρώπη και το αποτέλεσμα το βλέπουμε όλοι, μπροστά μας, στα μάτια μας. Οι εργαζόμενοι σήμερα είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του πληθυσμού που κινδυνεύει να βρεθεί κάτω από το όριο της φτώχειας. 10% των εργαζομένων αυτή τη στιγμή βρισκόνται κάτω από το ε, όριο αυτό. Και οι συντάξεις ε, των εργαζομένων είναι, που έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις είναι πάρα πολύ ψηλή, 8%. Λοιπόν, τι όριο θα δώσετε για αυτές τις καταστάσεις και άλλες διαθετικές μεταρρυθμίσεις, τι, μέχρι οι εργαζόμενοι να μην έχουν το νερό να πιούν, ναι. Αυτό περιμένουμε να μας πείτε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντομπρόφσκης να ξεκινήσει. Παρακαλώ. So uh, uh, ξεκινήσουμε από την πρώτη ερώτηση για την εφαρμογή των ειδικών συστάσεων αναχώρα. Όντως, ανησυχεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γεγονός ότι το ποσοστό εφαρμογής είναι σχετικά χαμηλό, ειδικά σε ό,τι αφορά την πλήρη εφαρμογή των ειδικών συστάσεων αναχώρα. Αλλά πιστεύουμε ότι ο τρόπος για να βελτιώσουμε την εφαρμογή είναι, περνάει μέσα από το διάλογο με τα κράτη-μέλη και μέσα από το διάλογο με τους ε, αρμόδιους φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους. Θέλω να τονίσω ακόμα ότι αυτές είναι συστάσεις, δεν είναι εντολές. Είναι συστάσεις σαν χώρα. Είναι κάτι που παράγει η Κομισιόν και που πιστεύει ότι διευκολύνει την ε, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ε, βελτίωση του κοινωνικού πλαισίου στα κράτη-μέλη. Είναι προς το συμφέρον λοιπόν των κρατών μελών να εφαρμόσουν επιτυχώς τις συστάσεις αυτές η Κομισιόν μπορεί να βοηθήσει. Απλώς. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία για να βελτιώσουμε την εφαρμογή μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των Ευρωπαϊκών Διαρθωτικών Ταμείων και Επενδυτικών Ταμείων Εδώ μιλάμε και για τη σωστή χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και μέσω της τεχνικής αρρωγής που μπορούμε να παράσχουμε στα κράτη-μέλη για την εφαρμογή των ειδικών συστάσεων αναχώρα μέσω της υπηρεσίας για την υποστήριξη των διαθωτικών μεταρρυθμίσεων. Πάω τώρα στην ερώτηση των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής. Δημοσιονομικά υπεύθυνες πολιτικές, διαθωτικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που γίνονται σε διάφορα κράτη-μέλη. Αυτές οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες πρέπει να αυξηθούν. Σε κάποιες χώρες όπως η Ιταλία ή η Γαλλία που αναφέρατε, έχουν γίνει σοβαρές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, ειδικά σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις για την αγορά εργασίας, το άνοιγμα κάποιων επαγγελμάτων, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς υπηρεσιών, παρότι σωστά είπατε ότι κάποιες από τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν απορρίφθηκαν σε δημοψήφισμα. Όμως είδαμε ότι υπάρχει πρόοδος στην ε, εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε αυτές τις χώρες. Σε ό,τι αφορά την έκθεση των πέντε προέδρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μία αξιολόγηση μάλλον διορθωνεμιλητή την Λευκή Βίβλο της Κομισιόν το Μάρτιο, όπου θα προτείνουμε τον τρόπο που θα προχωρήσουμε στην, ε, κεντρώνοντας στη δεύτερη φάση των όσων λέει η έκθεση των πέντε προέδρων. Γιατί η πρώτη φάση είτε έχει εφαρμοστεί ήδη ή είναι στη φάση με τους νομοθέτες. Ας πούμε έχουμε τώρα το Ευρωπαϊκό ε, Δημοσιονομικό Συμβούλιο, έχουμε το, τα Εθνικά Συμβούλια Παραγωγικότητας, ε, τις προτάσεις για την Τραπεζική Ένωση. Όλα αυτά τα έχουμε προτείνει πρόσφατα η Κομισιόν το ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων που έχει φτάσει στο επίπεδο των συνομοθετών κτλ. λοιπά. Για να πάω τώρα στα συγκεκριμένα ερωτήματα της Πορτογαλίας, με, με δημόσιο χρέος 130% ε, του ΑΕΠ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είναι σημαντικό να μειωθεί το έλλειμμα περιμένουμε ότι το έλλειμμα φέτος θα φτάσει στο 2,7 του ΑΕΠ και του χρόνου ε, θα φτάσει στο 2,3% του ΑΕΠ. Όμως, οι διαθωτικές μεταρρυθμίσεις ε, υπολείπονται σε σχέση με τις συστάσεις μας, γι' αυτό η αξιολόγηση που κάνουμε είναι ότι η Πορτογαλία αντιμετωπίζει κίνδυνο μη συμμόρφωσης. Ό,τι αφορά το ποσοστό ανάπτυξης, υπάρχει κάποια επιβράδυνση της ανάπτυξης ε, της Πορτογαλίας φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη και δυστυχώς ε, τα ποσοστά ανάπτυξης είναι σημαντικά κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επίτροπος Τάισεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα έλεγα ότι έχουν σε σχέση με τις απαντήσεις να προσθέσω ίσως κάτι εδώ για την Πορτογαλία η ανεργία είναι υψηλότερη από το μέσο όρο στην Πορτογαλία και έχουμε 10,8% πέρυσι ήταν 12,4% και η ανεργία των νέων στην Πορτογαλία είναι πολύ υψηλότερη από το μέσο όρο 28,9% τον Οκτώβριο φέτος και τον Οκτώβριο πέρυσι ήταν 32,1% είναι μια σημαντική μείωση αυτή που σημειώνεται λοιπόν στην ε, ανεργία και αυτό οφείλεται στο μεγάλο, στο μεγάλο ποσοστό στη μετανάστευση και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν τα ποσοστά της ανεργίας των νέων. Όμως αυτό πρέπει να το δούμε και σε σχέση και με άλλους συντελεστές. Για παράδειγμα, σε σχέση με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα κατά το οποίο σπουδάζουν ε, πολλοί νέοι και ασχολούνται με τις σπουδές τους και βλέπουμε ότι πάνω από 40.000 νέοι έχουν μετακινηθεί όσον αφορά το, τις δραστηριότητες ε, της ε, αντιμετώπισης ανεργίας των νέων και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τους νέους και όλα αυτά έχουν βοηθήσει να μειωθούν οι συντελεστές πρέπει να δούμε ότι διαφορετικά το ε, επίπεδο αυτό των 28 και παραπάνω της 100 δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Όμως ε, υπάρχει κάποια πρόοδος και ας συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστώ. Δύο λόγια για την Πορτογαλία να πω κι εγώ. Σωστό είναι ότι θεωρούμε πως η Πορτογαλία κινδυνεύει να μην συμμορφωθεί για τους λόγους που σας ανέφερε ο Βάλτης Ντομπρόφσκης. Παράλληλα όμως είπαμε ότι αυτή η κατηγορία είναι πολύ ετερογενής και είναι σε αρκετά καλή θέση αυτή την κατηγορία χωρών. Και αν επιβεβαιωθούν τα νούμερα που αναγγέλθηκαν, δεν θα χρειαστούν συμπληρωματικά μέτρα από την Πορτογαλία. Παρότι, όπως ακούσατε, ε, η διαρθρωτική προσπάθεια δεν είναι ακριβώς αυτή που ζητάμε. Υπολείπεται των αναγκών. Θα πρέπει να συνεχιστούν λοιπόν οι προσπάθειες, αλλά υπάρχουν και ενθαρρυντικά μηνύματα που δίνει η Πορτογαλία. Τέταρτος γύρος. Ένα λεπτό, ενάμιση λεπτό καθένας. Η κυρία Ζανόκα, από τους πράσινους. Ευχαριστώ την Επιτροπή που παρουσίασε κάποια θετικά αποτελέσματα. Ναι, ναι, βελτιώνεται το πράγμα αργά-αργά σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας. Αλλά όμως οι πιο φτωχές ε, περιφέρειες, και εγώ μια τέτοια εκπροσωπώ, ε, υποφελούνται λιγότερο από τα εργαλεία. Αυξάνεται, όπως ξέρετε, η φτώχεια. από αυτά που μας είπατε και από τα κείμενα που μας παρουσιάσατε, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν. Δεν βλέπω τίποτα καινούριο. Τα κλασικά που κοπανάτε κάθε φορά. Υπάρχουν και κάποιες ειδικέ συστάσεις βέβαια, παραδείγματος χάρη συγχρονισμός του κράτους πρόνοια, ούτω ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα για απασχόληση. Τι να καταλάβω από αυτό. Δηλαδή, να μειωθούν τόσο πολύ τα επιδόματα που οι άνεργοι θα πάρουν και θα δέχονται οποιαδήποτε δουλειά. Αυτό εννοείται. Θα ήθελα να θέσω μια συγκεκριμένη ερώτηση στην Επίτροπο Τάισεν, μια και δεν άκουσα ουσιαστική απάντηση στο ερώτημα που έθεσε ο εισηγητής μας για τα ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα. Και το ερώτημα είναι το εξή. Πότε θα παρουσιάσει η Κομισιόν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, μια οδηγία πλαίσιο για ένα ελάχιστο εισόδημα. Ευχαριστώ. κυρία Αγγέα, από το EFDD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπη. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρικ, ο οποίος αναφέρθηκε στην Ιταλία και στην, στο εντυπωσιακό αποτέλεσμα που πετύχαμε την περασμένη Κυριακή. Το 60% του Ιταλικού πληθυσμού συνεισέφερε για να διαφυλαχτεί το Σύνταγμά μας, που επί 68 χρόνια προστατεύει την ε, κυριαρχία και τη δημοκρατία της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν, γιατί νομίζω ότι η Ιταλία αποδεικνύει ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη θέληση του Ιταλικού λαού. Για τη σταθερότητα θα μιλήσουμε όταν δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να ψηφίσουν. Θα ήθελα να πω το εξή στους επιτρόπους τώρα. Είναι εύκολο να, να τα λέμε αυτά μεταξύ μας εδώ σε αυτόν τον οίκο. Εγώ θα ήθελα αυτά που μας είπατε σήμερα να τα πείτε στους πολίτες, σε όλους τους πολίτες και κυρίως στα 122 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που ζουν κάτω από το όριο φτώχεια και που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Γιατί το να μιλάτε για αυτή την θαυμάσια ευρωπαϊκή προσπάθεια, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπου όλοι είμαστε ευτυχισμένοι, όπου υπάρχει οικονομική ανάκαμψη, και μόνο τα ακούμε αυτά είναι ενοχλητικό, θα ήθελα να δω, να τα, να τα λέτε στου πολίτε και να δω και την αντίδρασή του, Γιατί ειλικρινά σα λέω. Θέλει, θέλει λιγάκι, θέλει πολύ θάρρο και διάθεση ας πούμε να αυτοτιμωρηθεί, για να πας να του τα πει αυτά. Δεν έχω να σα θέσω ερωτήματα. Ίσως εσείς θα πρέπει να μπείτε λιγάκι στην πραγματικότητα, να ξυπνήσετε εκεί πέρα και μόνο μετά από εκεί θα μπορέσετε να δώσετε συγκεκριμένες συνταγές βιώσιμες, πραγματικές για να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί ο ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους πολίτες που ζουν κάτω το ρίο της στόχιας περιμένουν αυτές τις λύσεις, αυτές τις συνταγές. Ο Μάρκο Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν υπάρχει περιθώριο για επιχειρηματολογίε εδώ. Φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει αντιληφθεί η ίδια την προβολική έλλειψη ισορροπία που έχει δημιουργήσει εντό τη Ευρωζώνη. Ιδίω ό,τι αφορά το εμπορικό ισοζύγιο κάποιων χωρών, μεταξύ των οποίων ακριβώ η Γερμανία. Το πιο σοβαρό είναι τη Ολλανδία. Και προτείνατε αυτή την δημοσιονομική επέκταση του 0,5% για 50 δις Αλλά για κάποιε χώρε όπω η Γερμανία και οι κάτω χώρε, η Ολλανδία, δεν θέλουν να το δεχτούν για λόγου πολιτικού. Ε, Πάντω από τεχνοκρατική πλευρά είναι συνεπή η στάση σα. Τουλάχιστον υπάρχει μια προσπάθεια να διαχειριστούμε αυτό που συμβαίνει. Βεβαίω, εδώ ήθελα να πω και κάτι πιο επιθετικό. Ήθελα να μου πείτε, εάν μπορείτε να δεσμευτείτε δημοσίω εδώ, ότι αν η Γερμανία δεν συμμορφωθεί με αυτέ τι συστάσει και μείνει σε αυτή την έλλειψη ισορροπία, μπορεί επιτέλου για πρώτη φορά να ανοίξει επί παραβάση τη δικασία εναντίον τη. Να κινηθεί τέτοια διαδικασία. Εδώ και 7 χρόνια έχουμε αυτό το πλεόνασμα που επαναλαμβάνεται. Ε, αυτό έχει κάνει μη βιώσιμη την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το νόμισμα ευρώ. Το 2016 κάποιοι που το υπέθεταν απλώς τώρα το βεβαιώνουν. Ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δημοσίω να λάβει θέση για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκίγκολτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μου φαίνεται λίγο τραγικό να σας ακούω διότι τρόπον τεινά οι διαπραγματεύσει, οι συστάσει που κάνατε προ το κράτη-μέλη, ιδίω στο πλαίσιο τη ετήσια έκθεση ανάπτυξη, δίνουν πολύ καλή, καλό υλικό ήδη. Ακόμη κι αν δυστυχώ η βιώσιμη μετάβαση στις αναχώρας τάση, έχει διαγραφεί σε σχέση με τις εκδοχές των προηγούμενων ετών. Όμως η πραγματική τραγωδία είναι που παρά την βραδύτατη πρόοδο, όπως εντόπισε και ο κύριος Χέκμαρκ, σε σχέση με την νομισματική πολιτική και τους προσανατολισμού της, παρά την βραδύτατη λοιπόν αυτή πρόοδο, δεν τολμάτε να πείτε ξεκάθαρα πόσο είναι ε, απογοητευτική αυτή η χαμηλότατη πρόσληψη των συστάσεων και των μεταρρυθμίσεων. Αν αυτού, ακούσουμε αυτό που είπε και ο κ. Σέκμαρ για τι συστάσει, ε, είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό υλοποίηση και χαμήλωσε τόσο πολύ από την αρχική φάση το 2012 που ήταν ήδη κακό. Οπότε, Επίτροπε Ντομπρόφσκη, αυτό δεν ισχύει απλώ για την πλήρη υλοποίηση μόνο. Ισχύει και για την ε, μερική υλοποίηση για αυτή την κατηγορία φαίνεται δηλαδή όλο ένα και περισσότερο να παραγνωρίζονται οι συστάσεις της Επιτροπής από τα κράτη. Η θαραλέα σας πρόταση για τη δημοσιονομική στάση απορρίφθηκε λίγο πολύ, για το δημοσιονομικό προσανατολισμό απορρίφθηκε λίγο πολύ απευθείας και ξεκάθαρα. Τι σκοπεύετε να κάνετε προκειμένου να βελτιώσετε την απόκριση των κρατών μελών. Ποια είναι η δική σας στρατηγική για να βρείτε κάποια λύση. Και επιτέλου ήθελα και μια σοβαρή απάντηση στην ερώτηση του κυρίου Χέκμαρκ. Οι καλοδεχούμενες βελτιώσεις από την πλευρά σας, ποιες βάσει των μακροοικονομικών σας μοντέλων θα είναι επιτυχημένες, μήπως θέλει η ακριβή δημοσιονομική πολιτική της ΕΚΤ, μήπως Πολύ μέρος από αυτή την πρόοδο είναι το αποτέλεσμα αυτής ακριβώς της πολιτικής της ΕΚΤ και τίποτε άλλο. Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα δεδομένα σας. Ναι, μπορείτε να μας προσχεθείτε να μην μιλάτε τόσο πολύ εκτός του χρόνου σας. Δεν θα προλάβουμε όλους τους ομιλητές αν το κάνετε αυτό. Η κυρία Κάπελ, ΕΝΕΦ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σε μείνω στα όρια του χρόνου. Έχω δύο ερωτήσει για τον Επίτροπο Ντομπρόφσκης σε σχέση με τις διαδοτικές μεταρρυθμίσεις και την προώθηση των ε, επενδύσεων και τον ε, ενάρετο, το ενάρετο αυτό τρίγωνο των επενδύσεων με την ανάπτυξη. Είπατε ότι έχουμε μέτρια ανάπτυξη, ότι πέφτουν τα ποσοστά ανεργίας, ότι το κρατικό χρέος μειώνεται και ότι τα ελλείμματα του προπολογισμού έχουν πάει κάτω από το 2% και το χρέος μειώνεται. Αυτό επιβεβαιώνεται από τι προβλέψει του φθινοπόρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ με το συμπεράσμά σα ότι αυτό δεν αρκεί. Και ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτουμε για να στρίξουμε την ανάπτυξη είναι η νομισματική πολιτική και τα χαμηλά επιτόκια τη ΕΚΤ. Όμω, κάποιοι λένε ότι η νομισματική πολιτική τη ΕΚΤ σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν λιγότερα κίνητρα να υλοποιήσουν τι διαφορετικέ του μεταρρυθμίσει. Διότι ακριβώ έχουν κρατική χρηματοδότηση και το πρόγραμμα αγορά ομολόγων το ενισχύει αυτό το, τελευταίο, το πρόγραμμα του τελευταίου χρόνου. Ιδίω για τι επενδυτικέ τράπεζε στον τραπεζικό τομέα υπάρχουν αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θέλω λοιπόν να μου πείτε εάν υπάρχει περίπτωση να γίνει εθνικοποίηση των τριών Ιταλικών τραπεζών, όπως έχει συζητηθεί. Ευχαριστούμε, Αντιπρόεδρος τον πρόφ. Ξεκινήστε. Ωραία. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. και πάλι για τις αναχώρα τάσεις και την υλοποίησή τους. Πρώτα απ' όλα είναι μία ε, ανησυχία που ε, και την Επιτροπή την απασχολεί και να πω ποιε είναι οι κατευθύνσει τι οποίες επεξεργαζόμαστε με τα κρατη μέλη για να υπάρξουν βελτιώσεις. Ε, μεταξύ των οποίων καλύτερο συντονισμό. και χρήση των κονδυλίων του ΕΦΣΙ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Ό,τι προσφέρουν τα διευθυντικά ταμεία, όλες οι μεταρρυθμίσεις που αναφέρονται στις αναχώρες συστάσεις και η δουλειά των κρατών μελών για να ετοιμάσουν τα δικά τους εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία να είναι περισσότερα συμμετοχικά, με μεγαλύτερη παρουσία των κοινωνικών εταίρων και των άλλων ενδιαφερομένων και για να ευαισθητοποιηθούν όλοι προς, ως προς τις προκλήσεις που είναι κοινέ και οι αποκρίσεις που θα πρέπει να πηχούνται στα εθνικά προγράμματα να, να μην είναι γνωστά μόνο σε μια υπηρεσία ενός Υπουργείου αλλά να είναι γνωστά γενικότερα στο επιτελείο ολόκληρου του κράτου, μέλους, του, ολόκληρου του κράτους που σχεδιάζει την πολιτική. Ως προς τα δεδομένα, τα συγκεκριμένα δεδομένα να απευθυνθείτε στους ειδικού. Και μόλις μας πούν και εμάς θα σας τα παράσχουμε. Ως προς το τους ενάρετους κύκλους ε, στην πολιτική της Γερμανίας και το πλεόνασμα. Ε, εδώ και ένα χρόνο έχει συζητηθεί το θέμα αυτό. Το πλεόνασμα θεωρείται ως μακροοικονομική έλλειψη ισορροπίας. Γι' αυτό η Γερμανία και κάτω χώρες λόγω χάρη θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες. Τους έχουμε απευθύνει σύσταση για να δούνε τι θα γίνει με τη ζήτηση στην οικονομία και τις επενδύσεις τους. Για την ΕΚΤ και την νομισματική πολιτική. Πρώτα απ' όλα, να θυμίσουμε ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ στοχεύει τον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός πρέπει να είναι κοντά ή κάτω από το 2%. Γι' αυτό ε, σχεδιάζεται έτσι η νομισματική της πολιτική, οπότε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούμε να σχολιάσουμε περιβολικά αυτές τις αποφάσεις της ΕΚΤ, πρέπει να σεβαστούμε για το δικό της κυρίαρχο δικαίωμα, την ανεξαρτησία της. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ένας από τους παράγοντες που κινητοποιούν την οικονομία. Όμως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν το χρόνο αυτό που έχουν για την νομισματική πολιτική για να περάσουν στις θετικές μεταρρυθμίσεις και να εκμεταλλευτούν το κενό. Ως προς τον τραπεζικό τομέα, αναφέρατε τις Ιταλικές τράπεζες, Είμαστε σε, διαρκές, σε, διαρκής, σε συνεχή επικοινωνία με τις Ιταλικές Αρχές και συζητούμε διάφορες λύσεις εντός του νομικού πλαισίου που διαθέτουμε αλλά και συγκεκριμένε επιμέρους τράπεζες δεν κάνουμε σχόλια. Ευχαριστούμε η κυρία Τάισον. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα σχολιάσω μόνο πολύ σύντομα το θέμα της φτώχειας και πάλι. Αν δει κανείς την κατάσταση στην Ευρώπη, θα δει κανείς ότι υπάρχει τεράστιος αριθμός διακυμάνσεων και διαφορών όσον αφορά τη φτώχεια το επίπεδο φτώχειας εκείνων που βρίσκονται υπό κίνδυνο αποκλεισμού και φτώχειας 13% έως 41% σε κάποια κρατημέλη. Μέσος όρος 23,7%. Όμως θα έλεγα όλα αυτά τα ποσοστά, ποσοστία μεγέθη, είτε είναι χαμηλά είτε υψηλά, εφόσον κάνουμε λόγο για ποσοστά φτώχειας, είναι πάντα υπερβολικά υψηλά. Κάνουμε λόγο για τη φτώχεια και κρύβονται πίσω από αυτού του αριθμού άνθρωποι και πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα τη φτώχεια. Τι κάνουμε. Έχουμε του στόχου τη στρατηγική 2020. Κατά τη διάρκεια τη κριση 2009 2009-2012 είδαμε να αυξάνονται τα ποσοστά φτώχεια και από τότε βλέπουμε ότι μειώνονται και βρισκόμαστε τώρα στα επίπεδα του 2009 και πάλι. Και πρέπει να πούμε ότι είναι ίσως χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με το 2008, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες, να συνεχίσουμε να έχουμε τα ορόσημα της στρατηγικής 2020. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην Ευρώπη είναι να παράσχουμε αρρωγή, να συνδράμουμε, να μπορέσουμε να παράσχουμε τη δυνατότητα και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και μέσω των κονδυλίων που θα διαθέσουμε. Το λέω αυτό σε σχέση με την εισήγηση και θα θυμούνται οι αρμόδιοι πόσο μεγάλη ήταν η μάχη που δόθηκε για να επιστρέψουμε επιστρέψουμε ώστε το 20% του ESF θα έπρεπε του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να διατίθεται προς αυτόν τον στόχο. Επίσης εργαζόμαστε σε σχέση με την καταπολέμηση της φτώχειας όσον αφορά τις συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Το κάνουμε αυτό ευθύ εξ αρχής από τότε που ξεκίνησε η προσπάθειά μας με οδηγίες και συστάσεις και έχουμε και συστάσεις ε, για την πολιτική όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας του 2008 βοηθούμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως ελάχιστον ελάχιστο μισθό μισθό. Υποστηρίζουμε το δίκτυο του ελάχιστου μισθού στην Ευρώπη και θα ήθελα να το τονίσω αυτό και να το υπογραμμίσω. Η φτώχεια είναι ένας τομέας που αφορά φυσικά κύρια και πρωταρχικά τα κράτη-μέλη. Μπορούμε να βοηθήσουμε εμεί, παρέχοντα ένα πλαίσιο, όμω είναι κυρίως πρωταρχικά το έργο των κρατών μελών να δράσουν και να αντιμετωπίσουν αυτή τη μάστιγα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν έτσι να δράσουν πιο αποτελεσματικά. Καμιά φορά δημιουργείται εντύπωση ότι η Ευρώπη μπορεί να επιλύσει όλα τα προβλήματα. Πολλά μπορούμε βέβαια να κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να εναρμονίσουμε τι διατάξει και του κανονισμού για την κοινωνική ασφάλιση και για να διασφαλίσουμε επίση τον ελάχιστο μισθό και όλες αυτές τις δράσεις που είναι αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των κρατών μελών. Και σε σχέση με, την, με το να κατηγορούμε γύροντας το δάχτυλο κατά της Ευρώπης δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας πιο αποτελεσματικά, στο πιο αποτελεσματικό επίπεδο εκάστοτε. Θα δράσουμε όμως από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να παροτρύνουμε και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να καταπολεμηθεί η φτώχεια. Ευχαριστώ. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Πάμε στον πέμπτο γύρο αποκρίσεων. Ενάμιση λεπτό έκαστο, το υπενθυμίζω. Ο κύριος Λένος από το ΕΛΚ είναι ο πρώτος μιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομος. Πολλά έχουν ακουστεί Θέλω να εστιάσω σε δύο συγκεκριμένα θέματα. Το πρώτο είναι η ανεργία των νέων. Όπω είπε πολύ σωστά η Επίτροπο ε, Τάισαν, υπάρχουν πάνω από 4 εκατομμύρια νέων ανέργων στην Ευρώπη σήμερα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια τέτοια κατάσταση. Είναι απαράδεκτη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για μια χαμένη γενιά νέων Ευρωπαίων, η σημερινή γενιά. Στην ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη του 2017, η Κομισιόν θα προτείνει μια νέα πρωτοβουλία για την νεολαία. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το θέμα και να μας πείτε από την εφαρμογή της εγγύησης για, την νέου, ε, για τους νέους και την ε, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για, του, τους νέους, τι διδάγματα μπορούμε να πάρουμε για αυτή τη νέα πρωτοβουλία. Γιατί φοβάμαι ότι επειδή η μάχη για την ενεργεία των νέων ε, πρέπει να δοθεί σε, σε επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο, ε, πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Επίση, α περάσουμε στου ηλικιωμένου. Έχουμε πολλέ βίβλου για τι συντάξει. Τη λευκή, την πράσινη κτλ. Βίβλου. Έχουμε κάνει πάρα πολλά για τι συντάξει. Ε, με στεναρότητα είπαμε ότι για να κρατήσουμε τι συντάξει σε βιώσιμο επίπεδο για το μέλλον θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στο δεύτερο πυλώνα, σε επικουρικές συντάξεις. Έχουμε λίγε τέτοιε στην Ευρώπη και διαρωτώ με πώ η Κομισιόν, πώ εμεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα για να δημιουργήσουμε περισσότερε τέτοιε επικουρικές συντάξεις σε επίπεδο κρατών μελών. Ευχαριστώ, κύριο Μπάλτ. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σχετικά σύντομο. Θα το προσπαθήσω. Ταυτόχρονα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μια σημαντική έκθεση μελέτη της ε, ε, Ένωσης του για την ε, εποπτεία των αγορών θα υπάρξουν τεράστια κονδύλια τα οποία ε, αποκρύπτονται από πλευρά των κρατών. Αυτό όσον αφορά και μια τεράστια μάζα, όσον αφορά ένα ανεδαφικό κοινωνικό σύστημα και μεγαλύτερες δαπάνες όσον αφορά την κατάσταση των προσφύγων που δεν μπορούν όλα αυτά να συνυπολογιστούν επαρκώς. Για παράδειγμα η δική μου χώρα, η Γερμανία, ήδη σε σχέση με το 2020 έχει τεράστιες δαπάνες όσον αφορά την χρέωσή της σε σημαντικό ε, ποσοστό και για το Λουξεμβούργο ε, έμεσα και ε, άμεσα δάνεια 22% ύψους και η Ολλανδία φτάνει ένα ποσοστό πάνω από 300% υπερχρέωσης βρίσκεται σε διαρκή απόσταση ε, σε σχέση με την αηφορία όσον αφορά αυτή την επιβάρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταλήγει όμως σε παρόμοια αποτελέσματα. Ερωτώ λοιπόν, δεδομένου του φόβου που δημιουργεί αυτή η κατάσταση όσον αφορά την υπερχρέωση, όσον αφορά τους ιδανικούς μαθητές, τους Γερμανούς, τώρα η προπαρασκευή όσον αφορά την ε, δημογραφική προσαρμογή που απαιτείται, μεγάλη μεταρρύθμιση ιδιαίτερα του συνταξιοδοτικού τομείου ή σε σχέση με τις δυνατότητες που πρέπει να εξευρεθούν. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροντρίγκες θα λάβει τώρα τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήμουν η συγγήτρια για αυτό το θέμα πέρσι και πρέπει να αναγνωρίσουμε το ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ των συστάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη νέα δέσμη μέτρων που παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Όταν, όσον αφορά το μείγμα πολιτικής με μεγαλύτερο βάρος για τις επενδύσεις, όσον αφορά τις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν, όμως θα ήθελα να επικεντρωθώ σε σχέση με τις συστάσεις που έγιναν διότι το γεγονός ότι υπάρχουν επιχειρήματα για τη συζήτηση όσον αφορά τα δημοσιονομικά και τα φορολογικά δείχνει ότι υφίσταται ένα πρόβλημα. Το αναγνωρίζει και η Ευρωομάδα σε σχέση με ένα χαρακτήρα οικονομικής μονάδας που έχει Ερώτησή μου, σε σχέση με αυτή τη μονάδα δεν θα έπρεπε να διοργανωθεί μια άλλη συζήτηση πώς μπορούμε να ανακτήσουμε και πάλι έναν θετικό κύκλο μέσα από αυτές τις προσπάθειες. Δηλαδή να μπορέσουμε όσον αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους, οικονομικούς στόχους και κοινωνικούς στόχους να μπορούμε να βαίνουμε εκ παραλίλου. Πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό αν δώσουμε το βάρος στην οικονομική και κοινωνική σύγκληση και συνοχή δίνοντας κίνητρα στα κράτη-μέλη να επενδύσουν επενδύσουν ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη ζήτηση και όλα αυτά θα δημιουργήσουν υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης σε όλον αυτόν τον κύκλο και θα καταστήσει ευκολότερο το να ε, επιτευχθεί η δημοσιονομική σταθεροποίηση και εξυγίανση. Αυτός ο γύρος θα έπρεπε, αυτός ο κύκλος θα έπρεπε να ακολουθηθεί νομίζω. Υπάρχει ένας όρος για να επιτευθεί αυτό, ότι όλα τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να έχουν μέσα και μέτρα για να επενδύσουν. Και πολλά δεν έχουν ή δεν υπάρχουν αυτά. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης. Ευχαριστώ για αυτό το θέμα της έμεσης χρέωσης στα πλαίσια και των δημογραφικών εξελίξεων. Αυτό που να ληφθεί υπόψη ιδίως ό,τι αφορά την μακρόπνοη βιωσιμότητα των, του συστήματος των συντάξεων και κοινωνικών ασφαλίσεων. Αυτό το έχουμε ήδη εξετάσει στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μέσω των ειδικών συστάσεων αναχώρα, μέσω της διασύνδεσης της ε, συνταξιδοτικής ηλικία με το προσδόκιμο ζωής, του συνταξιδοτικού ορίου δηλαδή με το προσδόκιμο ζωής και μέσω άλλων μεταρρυθμίσεων στις συντάξεις, ούτως ώστε να βελτιώσουμε την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων των μας. Όσο λιγότερες διορθώσεις κάνουμε, γιατί ενσωματώνουμε τις τάσεις και τις, και τις βελτιώνουμε, τόσο λιγότερες αυτό το καλύτερο. Ε, είναι ένα μακρόπνο θέμα που απαιτεί συνεχή προετοιμασία και δουλειά. Τώρα για τις συστάσεις της Ευρωζώνης και τις προτεραιότητες της σύγκλησης των επενδύσεων, της μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό ευθυγραμμίζεται και συνδέεται με τις με τα μεγάλα προβλήματα, με μεγάλες ανησυχίες κομισιών, ε, πρέπει να υπάρξει σύγκληση προς τα πάνω και αυτό το λέει όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά το λέμε και στις προτάσεις μας για την ολοκλήρωση της ε, Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Και θα συνεχίσουμε και, στην, και με τη δεύτερη φάση της έκθεσης των πέντε προέδρων να το κάνουμε προτεραιότητα. Ήταν προτεραιότητα δηλαδή από την αρχή που ανέλαβε αυτή η Κομισιόν τα καθήκοντά της. Η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων είναι κάτι που μας απασχολεί και θα μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο στο φετινό Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, όπως απεικονίζεται και στην ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ, Επίτροπο Τάισεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα για την πρωτοβουλία για τους νέους. Υπήρξε ερώτηση σχετικά και θα ήθελα να τοποθετηθώ. Εμείς προτείναμε κάποιες μέρες ε, πριν, πολύ πρόσφατα, και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να γίνουν περισσότερα για τους νέους. Δεν θέλαμε αυτή η γενεά να μείνει πίσω και να χωλένει και θέλαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Ρωτήσατε τι γίνεται σε σχέση με την πρωτοβουλία απασχόληση των νέων και ποια αποτελέσματα παράγονται. Μειώνεται η ανεργία των νέων και το είδαμε αυτό. Κάνουμε λόγο για μια διαθωτική μεταρρύθμιση και θα δούμε τα αποτελέσματα μελλοντικά βέβαια. Αλλά πρέπει να επενδυθούν περισσότερα κονδύλια σε αυτή την προσπάθεια. Γι' αυτό και μέρος αυτών των κονδυλίων και μέρος αυτής της πρότασης, δηλαδή ένα δις ευρώ να προσθεθεί στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και όλα αυτά θα ακολουθηθούν και από ένα πρόσθετο ακόμα δις ώστε τα κράτη-μέλη που, που εξακολουθούν και πλήττονται από υψηλότατα ποσοστά ανεργίας νέων θα τύχουν συνδρομής μέσω αυτών των κονδυλίων. Ένας άλλος τομέας μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη, τα ειδικά μέτρα που προτείναμε και με την πρόταση για την επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση που έχουμε καταθέσει ώστε να μπορέσει η διτή εκπαίδευση να διασφαλιστεί, dual training, να υπάρχει δυνατότητα μάθησης επιτόπου και να μπορέσουμε διασυνοριακά να προχωρήσουμε στην ε, απόκτηση αυτών των ε, δεξιοτήτων. Ένα πρόγραμμα Erasmus Sin, Erasmus Plus, ώστε να μπορέσουν ε, να συνδυαστούν αυτοί οι στόχοι όσον αφορά και την κατάρτιση για να υποφεληθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα οι υποφελούμενοι, να μπορούν από έξι μήνες έως ένα έτος να μεταβαίνουν στο εξωτερικό στην Αλοδαπή. Εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας φυσικά, αυτό συνεισφέρει μέσω αυτών των προτάσεων και έτσι να υπάρχει και το εθελοντικό σώμα υπηρεσίας ώστε οι νέοι να συμμετέχουν και να έχουν κίνητρα να συμμετάσχουν στο ε, σώμα εθελοντών για να μπορέσουν να δράσουν ε, ε, και να συνδράμουν στο εξωτερικό με την εθελοντική τους εργασία. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα. Εκεί αυτή απουσιάζει και μέσω της εθελοντικής υπηρεσίας μπορούν να καλύψουν αυτά τα κενά, μπορούν να εκμάθουν μια γλώσσα, μπορούν να αποκτήσουν τα, τις και την κατάρτιση ώστε να μάθουν κάποιο επάγγελμα, πράγματα τα οποία, ένα επάγγελμα, ε, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να μάθει κανείς σε ένα σχολείο. Παράδειγμα, ε, επαγγελματικά να μπορέσουν να καταρτιστούν και να αποκτήσουν πείρα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει αναπτύξουμε περαιτέρω αναπτύσσοντας τον τρίτο πυλώνα περισσότερο βλέποντας ότι έχει αναπτυχθεί ο δεύτερος περισσότερο να δώσουμε μέτρα ώστε να υποφεληθούν οι νέοι από αυτά. Να απαντήσω με δύο λόγια στην κυρία Ροντρίγκε. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι υπάρχουν κάποιοι διεθνεί οργανισμοί, το G20 ή το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο ή ο ΣΑ, που θεωρούν ότι σε περίπτωση πολύ ασθενούς ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουμε όλους τους κινητήρες της ανάπτυξης. Την οικονομική πολιτική, παρότι πρέπει να κάνουμε τις ε, προσαρμογές, τις απαραίτητες προσαρμογές. Το σχέδιο Juncker για τις επενδύσεις, το οποίο το ενισχύσαμε και το παρατείναμε το παρατείνομαι. 500 εκατομμύρια, 500 ε, δισεκατομμύρια συγγνώμη, ευρώ μέχρι το 2020. Επίσης, ε, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις ε, για το ανθρώπινο κεφάλαιο, εκπαίδευση κτλ. Και το υπόλοιπο τι είναι, δημοσιονομικές πολιτικές. Τι διαπιστώνουμε γι' αυτό. Υπάρχει μια δημοσιονομική εξυγίαση που έδωσε πολύ ωραία αποτελέσματα. 1,5% και ουδέτερος δημοσιονομικός προσανατολισμός σήμερα. Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε το δυναμικό ανάπτυξη Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει επίσης να έχουμε μια θετική ε, δημοσιονομική, ε, δημοσιονομικό άθροισμα. Το 0,5% δεν το ήθελε αυτό η Κομισιόν. Η Κομισιόν ήθελε να, γίνει, να τεθεί το θέμα και να αναγνωρίσουμε την ανάγκη ενός δημοσιονομικού ε, διαφόρων δημοσιονομικών κινήτρων και να μειωθούν οι ανισορροπίες που υπάρχουν, οι... τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα. Έγινε μια πρώτη συζήτηση λοιπόν στο Eurogroup και αναγνώρισε τουλάχιστον ότι είναι σωστή η προσέγγιση της Κομισιόν. Θεωρώ, θετικό είναι. Εν συνεχεία θα δούμε και τα συμπεράσματα. Όπως είπε και ο Γερούν Ντάισερ Μπλουμ, ε, είμαστε σε μια φάση μεταβατική. Και σε αυτή την ε, μετάβαση χρειαζόμαστε ε, μια νέα τροχία για τις οικονομικές πολιτικές. Ευχαριστώ. Εάν μου επιτρέπετε να δώσω μια τελευταία φορά σε έναν την ευκαιρία στην κυρία Μωρά Σαρτιέ που θέλει να μας μιλήσει για το κοινωνικό ταμείο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, να με συγχωρούν οι Επιτροποί. Δυστυχώς ε, βρισκόμαστε στο Προεδρείο του Κοινοβουλίου, γι' αυτό ακριβώς καθυστέρησα. Αλλά όχι από έλλειψη ενδιαφέροντος. Ήθελα να σχολιάσω την κοινή βούληση όλων να αντιμετωπίσουμε τι κοινωνικέ ανισορροπίε με την εργασία, την ένταξη στην αγορά εργασία. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των νέων χωρί προσόντα για να ενταχθούν στην αγορά εργασία, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να προσέξουμε και κάποιε ομάδε του πληθυσμού που είναι ευάλωτε, όπω οι γυναίκε, οι οποίε πετάχτηκαν από την αγορά εργασία λόγω τη κρίση και θα πρέπει να ανταποκριθούμε πολύ γρήγορα και στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ωστόσο, δεν αναγκαζόμαστε να βοηθούμε έτσι τα κρατημέλη να αλλάξουν αυτήν την ίδια την αντίληψη της εκπαίδευσης, της κατάρτισης. Για την ώρα είμαστε προσανατολισμένοι στο εκπαιδευτικό σύστημα που δίνει πτυχία. Κρατάνε περισσότερο αυτές τις διαδικασίες. Δεν πρέπει σήμερα να δραστηριοποιήσουμε πολύ πιο έντονα την αναγνώριση των δεξιοτήτων, δεξιοτήτων που θα επιτρέπει μεγαλύτερη κινητικότητα, μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και προσαρμογή στι ανάγκε των επιχειρήσεων και μεγαλύτερη κυκλοφορία, για να μην πω πλούτο ε, για τα βιογραφικά των ανθρώπων, ώστε με την αναγνώριση δεξιοτήτων τους, δεξιοτήτων που έχουν ε, αποκτηθεί εκτός επαγγελματικού χώρου, έρχομαι σε αυτό που είπε η Επίτροπος Τάισεν για τους εθελοντές στο σώμα αλληλεγγύης, οι νέοι αυτοί θα αποκτήσουν δεξιότητες. Θα πρέπει αυτές οι δεξιότητες, αυτά τα προσόντα να αναγνωριστούν και να συμπεριληφθούν σε ένα δέντρο δεξιοτήτων το ίδιο και οι γυναίκες. Πολλές φορές έχουν ε, επενδύσει και ασχοληθεί σε συλλόγους, σε ενώσεις. Πρέπει και αυτές μέσω αυτής της αναγνώρισης των δεξιοτήτων να ε, ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και ένα εργαλείο για να το πετύχουμε αυτό είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Thank you. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ όλους σας για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ όμως τους Επιτρόπους, τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκης, την Επίτροπο Τάισεν και τον Επίτροπο Μοσχοβησή. Ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν είχαμε όμως κάποιο λαβράκι ε, να ακούσουμε σαφή στοιχεία και αριθμούς και πολύ σοβαρά επιχειρήματα από όλες τις πλευρές. Σας ευχαριστώ πολύ.